Καλημέρα. Καλώς ήρθατε ε, στο κοινό μας εργαστήριο με την Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, σχετικά με, τις, ε, με τους οργανισμούς Καθώ επίσης ε, συγκεκριμένα για την υποπτία και πόρη εν μέρει και πλήρω αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών. Ε, το ζήτημα που μας αφορά είναι οι απαλλαγέ ε, και ιδιαιτέρω για αυτούς τους οργανισμούς που έχουν, επιτελούν έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως ε, να ε, συμμετέχουν στον προϋπολογισμό. Θα θέλαμε να ε, καλωσορίσουμε τον κύριο Γκάια και Βόγκαν, ο οποίος όμως εκπροσωπείται από την κυρία Μάια, η οποία στη συνέχεια θα αναλάβει και την Προεδρία εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, καθώς επίσης και τους προσώπους της Κομισιόν από το δίκτυο των ε, οργανισμών ε, έχουμε τον κύριο ε, Σπανιόλη από την ΕΦΣΑ, την καθηγήτρια Βος από το Academic Research Network on Agentification of EU e Executive Governance, το TARN, την Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, επίσης ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ΕΚΒΑΤ ε, από, την αυτοχρηματοδοτούμενο, από αυτοχρηματοδοτούμενο οργανισμό καθώς επίσης και τον κύριο Μάστιο από την ΑΣΑ ε, εσείς είσαστε επίσης υπεύθυνο για την ευελιξία των ε, πόρων ε, και όλο αυτό μας ενδιαφέρει. Έχετε τη δυνατότητα 10 με 15 λεπτά να μιλήσετε. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε ανάμεσά μας και ανυπομονούμε να ακούσουμε τις παρουσιάσεις σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον γνωμοδότη. Ευχαριστώ, Ίνκε. Ε, δυστυχώς ο κύριος Κάιερ ε, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, ε, όμως περιμένουμε τη Μόνικα Χελμάια από την Επιτροπή Προπολογισμών. Σε λίγο, ίσως μέχρι να έχω τελειώσει θα έχει έρθει και θα μπορέσει να πει και αυτή κάτι γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ε, για, τις, ε, ε, για τους οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται είτε από αμοιβέ, είτε χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα τον γνωμοδότη για τις απαλλαγές. Πρότεινα στο γνωμοδότη να έχουμε ένα κοινό εργαστήριο. Βλέπουμε ότι έχουν έρθει πάρα πολύ σήμερα ε, ίσως ε, από τις ε, μεγαλύτερες, από τις λίγες φορές που έχουμε τόσους πολλούς προσκεκλημένους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σε αυτό το εργαστήριο και ευελπιστώ να σας φανεί ενδιαφέρον. Θα ήθελα να προτείνω πρότεινα μάλλον το συγκεκριμένο εργαστήριο για διάφορους λόγους είναι λοιπόν μια ευκαιρία αφενός να εξετάσουμε το πώς θα ορίζουμε τις αμοιβέ, πώς οι υπηρεσίες αυτές θα γίνονται και αν είναι χρήσιμο ε, να συμπεριλαμβάνουμε και ε, πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς στη διαδικασία απαλλαγής. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι οργανισμοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται από ε, αμοιβέ ασκούν μικρότερη πίεση στον προπολογισμό της Ένωσης διότι όπως γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο μεγάλος όσο θα ήθελαν ε, μερικοί ε, ιδιαίτερο όσον αφορά ας πούμε, την πολιτική συνεχή. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει μεγάλη πίεση στον προπολογισμό τη Ένωση σε περίπτωση που υπάρχουν αμοιβέ για αυτέ τι υπηρεσίε. Επίσης, όταν συζητήσαμε για τις απαλλαγές, ε, μιλήσαμε, μιλήσαμε πολύ και για τις ε, μεταφορές ε, στους προϋπολογισμούς. υπάρχουν ακόμα οργανισμοί οι οποίοι κάνουν μεταφορές στο τέλος του οικονομικού έτους όμως αυτές οι μεταφορές μπορεί να είναι χρήσιμες ε, για να αντιμετωπιστούν ε, ξαφνικά γεγονότα ε, και πράγματι χρησιμοποιώντας αυτές τις μεταφορές έχουμε τη δυνατότητα της ευελιξίας για, τις, για τους οργανισμούς ούτως ώστε να λάβουν δράση σε περίπτωση που συμβεί κάτι ξαφνικό. Ε, παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ε, στην σύγκρουση συμφερόντων ε, όταν υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί μεταξύ των οργανισμών αλλά και της οικονομικής εξάρτησης από τις βιομηχανίες, Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ορθή ισορροπία και θα πρέπει να παρακολουθούμε και τις σχέσεις που έχουν οι βιομηχανίες με αυτούς τους οργανισμούς με βάση το συγκεκριμένο, τη, τη σημερινή εκδήλωση θα ήθελα ε, να γύρω κάποια ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να έχουμε διάφορες απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα ποιος ορίζει τις αμοιβέ, πώς ε, καθορίζονται, ε, πώς, αν θα πρέπει να ορίζονται από, τη, από οικονομικούς κανονισμούς, αν τα πλεονάσματα τα οποία προκύπτουν θα πρέπει να κρατώνται και τι να γίνονται, πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, πού μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτά τα πλεονάσματα, αν θα πρέπει να, ε, να, να προστίθενται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ε, αν θα πρέπει ε, να ε, συμμετέχουν στη διαδικασία απαλλαγής οι συγκεκριμένοι οργανισμοί αν θα πρέπει οι συγκεκριμένοι οργανισμοί να ε, έχουν τις ίδιες περικοπές προσωπικού όπως έχουν και άλλοι οργανισμοί ε, για ε, εξοικονόμηση πόρων εφόσον τα χρήματα δεν προέρχονται από τον προπολογισμό της Ένωσης ακούμε διαμαρτυρίες κάθε χρόνο και όσον αφορά το, τη μείωση του 5% αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν και ε, στην μεταφορά προσωπικού. Έτσι λοιπόν, αν θα πρέπει ε, να συμμετέχουν σε αυτή τη μείωση προσωπικού και στην απλοποίηση της διαδικασίας. Ε, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν σήμερα. Δεν ξέρω αν θα λάβουμε απαντήσεις για όλα αυτά, όμως τουλάχιστον θα είναι ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε όλα αυτά, ούτως ώστε να υπάρξει μια διάβγεια πάνω σε όλα αυτά και στο μέλλον θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τι απαραίτητε αλλαγέ Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, πολύ. Μόλις ήρθε η συμπροεδρεύουσα, η κυρία Μάγια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια πρώτα ε, σχόλια. Ε, με τα οποία ασχολείται και η Κομισιόν εδώ και καιρό. Αρχικά όσον αφορά τις συζητήσεις με τους οργανισμούς είναι ε, δύσκολο με αυτήν την ε, διαδικασία ε, μεταφοράς προσωπικού. Είναι μια πολύ τεχνοκρατική διαδικασία και γι' αυτό το λόγο είμαστε ιδιαίτερα κριτικοί. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό project, όμως παρατηρούμε και μια τάση να μην έχουμε υπόψη μας τις αμοιβέ ε, βλέπουμε δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν πολύ εύκολα να πληρώσουν αυτές τις αμοιβέ ε, και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να υπάρξει μια, ένας μηχανισμός για την αλλαγή της δομής των αμοιβών. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δεν είναι ευέλικτο και δεν είναι ανάλογο της κατάστασης των διαφόρων οργανισμών. Το μοντέλο της ΕΑΣΑ για παράδειγμα το βρίσκω πολύ καλό διότι βραχυπρόθεσμα ε, αποφεύγει αυτές τις διακυμάνσεις ε, προσωπικού ε, και υπάρχει και μια επιπρόσθετη ε, διαδικασία ελέγχου ε, σχετικά με, το, με τα νέα πρότυπα τα οποία εισάγονται, όποτε προστίθεται μια τεχνολογία για παράδειγμα, τότε έχουμε νέες αιτήσει, όμως στη συνέχεια έχουμε λιγότερες αιτήσει, διότι η, ο φόρτος εργασίας έχει μειωθεί ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι πάνω σε αυτό και ε, το θεωρώ θετικό το γεγονός ότι λαμβάνουμε υπόψη μας ε, και τις αμοιβέ οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και οι, ίδιες, οι ίδιοι οργανισμοί θα, θα μπορούν να είναι πιο ευέλικτοι σε ό,τι και αν προκύπτει. Θα ήθελα Προσφάτως αναφέρθηκε μια, ε, ένα παράδειγμα στην ΕΦΣΑ η οποία έπρεπε να επεξεργαστεί πάνω από 150 αιτήσει ε, ε, βλέπουμε ε, λοιπόν ότι ε, ξαφνικά ενώ περίμεναν για παράδειγμα 150-200 αιτήσει είχαν χίλιες αιτήσει να επεξεργαστούν. Αυτό λοιπόν όσον αφορά, αυτό όσον αφορά την ευελιξία λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Ταυτόχρονα όμως οι αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί το θέμα το οποίο γύρεται, όπως λέει ο κύριος Γκάιερ, είναι ε, το ζήτημα της ανεξαρτησίας, ε, διότι μπορεί να επηρεάζονται οι οργανισμοί αυτοί από τις, ε, στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις επειδή έχουν συνεισφέρει οικονομικά σε μεγάλο βαθμό. Ε, το πιλωτικό πρόγραμμα της ε, ΆΣΑ είπε ότι αποτελεί μια καλή ε, βάση, μας ικανοποιεί και συμφωνώ με αυτό. Ε, βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, σε όλους τους οργανισμούς, ούτε η τεχνοκρατική διαδικασία, ώστε να πούμε ότι λειτουργεί στην ΕΑΣΑ σημαίνει ότι θα είναι καλό ε, και για οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, διότι συγκεκριμένα θα πρέπει να συζητήσουμε με τους οργανισμούς και να εξετάσουμε μονομένες δυνατότητες που υπάρχουν για την βελτίωση του εκάστοτε οργανισμού. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω προσωπικό, προσωπικά είναι ότι όταν έχουμε πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, τότε τα χρήματα τα οποία έχουν αυτοί οι οργανισμοί δεν μπορούν να εξαφανίζονται στο γενικό προϋπολογισμό, είτε θα μειωθούν οι αμοιβέ, ούτω ώστε να μην ε, έχουν αυτοί οι οργανισμοί πολλά χρήματα. Ε, Ιδάλλως ε, θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό μοντέλο σχετικά με το πώς ε, θα μπορούμε να απαλλάσσουμε άλλους οργανισμούς ε, αλλά το να κρατάμε ε, ποσά ε, όπως είναι για παράδειγμα διάφορους οργανισμούς αυτό δεν είναι σωστό εφόσον λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που δεν χρειάζονται μεγάλο αριθμό προσωπικού τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχουν μεγάλες αμαβές θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαλεία ανάλογα με, την, τον οργανισμό και ανάλογα να προσαρμόζονται οι διάφορες αμοιβέ. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς, ε, είστε ακριβώς στο επίκεντρο του θέματος ε, και περνάμε στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Σιλβάνο Πρέσα από την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και την κυρία Ο σκοπός της παρουσίας μου, παρουσίασής μου σήμερα είναι να σας δώσω μία επισκόπηση, κάτι το οποίο σε έναν βαθμό έχει κάνει ε, ο και να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές ε, της σημερινής ε, παρουσίασης που είναι η εποπτεία και η πόρη. Δύο θέματα λοιπόν θα με απασχολήσουν ιδιαίτερως ε, σήμερα. Είναι αρχικά το πώς διαχειριζόμαστε τα έσοδα από αυτά τα τέλη, αυτές τις αμοιβέ και δεύτερον το ανθρώπινο δυναμικό ο αριθμός των υπαλλήλων σε αυτούς τους οργανισμούς. Και εδώ βεβαίως υπάρχει διασύνδεση και με τον γενικότερο στόχο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την τρέχουσα περίοδο, να υπάρχει μια συνολική μείωση του αριθμού των, ε, του προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων κατά 5% αλλά και ε, στις ε, υπηρεσίες και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Υπάρχει όμως και ένα αίτημα παράλληλα που ανέφεραν οι προηγούμενοι μιλητέ ότι οι οργανισμοί που βασίζονται σε έσοδα από τέλη θα πρέπει να τα και στις, ε, στα αιτήματα της αγοράς, στις ανάγκες της αγοράς, ε, να ανταποκριθούν ε, σε διακυμάνσεις, στο φόρτο και στις ε, συνθήκες της αγοράς. Τώρα, αυτοί οι οργανισμοί που βασίζονται σε έσοδα από τέλη, πόσοι είναι και αν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Συνολικά, Έχουμε 8 τέτοιους οργανισμούς, είτε μερικώς είτε πλήρως χρηματοδοτούμενοι από αυτά τα τέλη. Έχουμε τρεις αποκεντρωμένους οργανισμούς που εν μέρη χρηματοδοτούνται από τέλη που καταβάλει ο κλάδος, ε, συγκεκριμένα ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας και ο Ευρωπαϊκός ε, Οργανισμός Χημίας, που εδώ έχει διάφορα τμήματα βέβαια, μπορούμε να τα δούμε όλα από κοινού. Μετά έχουμε μια δεύτερη κατηγορία που χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό και εν μέρη από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι οι τρεις εποπτικές ε, ε, αρχές των χρηματοοικονομικών που είναι η Ευρωπαϊκή ε, η EBA, Security and Markets Authority. Τέλος έχουμε δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που καλύπτονται από ε, τον κλάδο, το Γραφείο Δικαιωμάτων ε, Γενοτικής Ιδιοκτησίας και τέλος το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών ποικιλίων. Επομένω, ακόμα και στο πλαίσιο των ε, οργανισμών που βασίζονται σε έσοδα αποτέλει, έχουμε διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότηση και διάφοροι φορεί ε, εμπλέκονται ε, στα έσοδα που συλλέγονται από αυτούς τους οργανισμούς. Τώρα, πώς έχει η διαχείριση των εσόδων αυτών αποτέλει. Έχουμε δύο βασικά μοντέλα Έχουμε οργανισμούς όπου όλες ε, οι πηγές ε, εσόδων ε, την χάνουν της ίδιας διαχείρισης από κοινού. Είναι λοιπόν ένα εισόδημα για τους οργανισμούς με το οποίο μπορούν να καλύψουν όλες τις δαπάνες τους. Μετά έχουμε και ένα δεύτερο μοντέλο όπου οι διάφορες δραστηριότητες των οργανισμών διαφοροποιούνται και τα έσοδα αποτελεί ουσιαστικά καλύπτουν δραστηριότητες που έχουν άμεση συνάφεια με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός. Στην πράξη και τα δύο μοντέλα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν καλά, έχουν διαφορές βεβαίως. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ε, μοντέλο που όλα τα έσοδα καλύπτουν όλες τις δαπάνες έχει χαμηλότερο διοικητικό άχθος και περιορίζει ε, την διαμόρφωση μεγάλων αποθεματικών που να προκύπτουν από τέτοια έσοδα αποτέλη τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι όταν έχουμε αποθεματικά στον ε, ετήσιο προπολογισμό των οργανισμών, εκεί υπάρχει η δυνατότητα ε, να μεταφερθεί ως ε, εισόδημα για ειδικό προορισμό και σε κάποιες περιπτώσεις έχει οδηγήσει αυτό στη δημιουργία σημαντικών αποθεματικών που είναι και το χαρακτηριστικό ορισμένο από αυτών των οργανισμών. Τώρα, Ας περάσω στο δεύτερο σκέλος αυτών των πόρων που, ε, των πόρων που μετρώνται σε όρους εξέλιξης ε, του προσωπικού. Δηλαδή ο αριθμός ε, των θέσεων που επιτρέπονται στο σχέδιο απασχολησιμότητας αυτών των οργανισμών. Εδώ στο γράφημα βλέπετε την εξέλιξη από το 2007 μέχρι το 2017 μπορείτε να δείτε ότι μέχρι τα 2013 είχαμε μια σαφή αυξητική τάση σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Εν μέρει αυτό ε, προέκυψε από το γεγονός ότι αυξήθηκε ο ρυθμός στον οργανισμό. Το 2010 είχαμε την ε, ε, δημιουργία των τριών εποπτικών αρχών, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη η αύξηση. Από το 2013 και μετά και μετά τη συμφωνία για να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός ε, των υπαλλήλων Βλέπουμε λοιπόν μια σταθεροποίηση και έτσι άλλαξε και η τάση. που συνδέεται στενά με την ε, δημοσιονομική εποπτεία και για αυτούς τους οργανισμούς και για τους υπόλοιπους βεβαίως σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ανθρωπινών πόρων. Το 2013 θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση όπου παρουσίασε ένα ε, προγραμματισμό των ε, ε, επιπέδων ανθρωπινών πόρων των οργανισμών και μεμονωμένα και συνολικά και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε στην μείωση του προσωπικού κατά 5%. Από τότε είχαμε διάφορες αποφάσεις που ελήφθησαν στις αιτήσει δημοσιονομικές διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε διάφορες περιπτώσεις βέβαια έχουν αποφασίσει να αποκλει... παρεκκλίνουν αυτής της, ε, αυτού του στόχου για τους ανθρώπινους πόρους. Συνολικά, εξετάζοντας ε, και το σχεδιασμό στον ετήσιο προπολογισμό, μεταξύ του 13 και του 17 έχουμε μείωση της τάξης του 1,8%, που είναι χαμηλότερη από τον στόχο, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι αλλάζει ε, η γενικότερη τάση. Αυτό που ανέφερε και ο κύριος Βον και η κυρία Χολμάιερ, τι κάνουμε όταν αλλάζουν οι απαιτήσει της αγοράς. Αναγνωρίζουμε ότι εδώ για, τις, για τους οργανισμούς που βασίζονται σε τέλη, ε, υπάρχουν ορισμένε μεταβλητέ, και έτσι υπάρχει μια εξάρτηση από την αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο ε, της ε, διοργανικής ομάδας εργασίας για τους Ευρωπαϊκού οργανισμούς υπήρξε μια συζήτηση να έχουμε μια διαφοροποιημένη μεταχείριση για τους ε, οργανισμούς που βασίζονται στα τέλη και να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό έργο το οποίο ε, εφαρμόστηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και ε, αυτό το πιλωτικό έργο ουσιαστικά ήθελε να εντοπίσει ορισμένους ε, σημαντικούς και χρήσιμους δείκτες φόρτου εργασίας και απόδοσης που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς ε, για να αποφασίσουμε τα επίπεδα ε, προσωπικού που θα πρέπει να έχει ο κάθε οργανισμός και έτσι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μεταβολές και διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτό βέβαια είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ή μάλλον και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Είδαμε ότι ε, τα σημερινά επίπεδα τελών είναι τα κατάλληλα. Υποθέσαμε λοιπόν ότι τα επίπεδα ήταν τα κατάλληλα και η προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των δικτών είναι η ύπαρξη ε, μηχανισμών, ελεγκτικών μηχανισμών που μας ε, επιτρέπουν να έχουμε αξιόπιστους ε, και χρήσιμους δείκτες. Στοχός ήταν αυτοί οι δείκτες κατά την κατάρτιση του υπερπολογισμού και της έγκρισης του να προσαρμόσουμε τα επίπεδα ανθρωπίνων πόρων των οργανισμών ανάλογα με τις ε, αναμενόμενες αλλαγές ε, στη ζήτηση. Υπήρξε λοιπόν η υπόθεση ότι αλλαγές ε, στους δείκτες, στο φόρτο εργασίας μέσα σε ένα εύρος συν πλην 2% μπορούν να θεωρηθούν μια φυσιολογική εξέλιξη και δεν απαιτούν ε, τροποποίηση των επιπέδων ανθρωπίνων πόρων. Όταν όμως ε, οι διακυμάνσεις είναι μεγαλύτερες, πάνω από το σύμπλην 2%, εκεί θα πρέπει να αλλάξουμε και τα επίπεδα του προσωπικού. Αυτό ελέγχθηκε πρώτη φορά στον προπολογισμό του 2017 και αντί να έχουμε τελικά πτώση ε, του αριθμού των υπαλλήλων ε, της ΕΑΖΑ, ουσιαστικά σταθεροποιήθηκε ο αριθμός και χρησιμοποιήσαμε τον δίκτυο αυτό ως μία αναφοράς. Αυτό το πιλωτικό έργο ε, συζητήθηκε και στη διοργανική ομάδα Εργασίας από πλευράς Κοινοβουλίου ήταν μάλλον ενθαρρυντική η υποδοχή. Από την πλευρά του Συμβουλίου υπάρχει μια επιφύλαξη για να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως ε, μοντέλο, σημείο αναφοράς για την κατανομή των πόρων. Μας είπαν ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι αυτός που μετράει και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Εμείς βέβαια θέλουμε κάπως να συγκεράσουμε αυτές τις ε, διαφορετικές απόψεις. Κλείνοντας, να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς συζήτηση, τα οποία ανέφεραν και οι Εδώ θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να βρουν τη σωστή ε, ισορροπία με μια κατάλληλη και σωστή χρήση των πόρων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετά κατά πόσο μπορούμε, μπορούν τα θεσμικά όργανα να αποφύγουν, να αποποιηθούν την ευθύνη ε, για την εποπτεία και τον έλεγχο. Αυτό ισχύει για τις πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενες ε, υπηρεσίες που δεν έχουν αντίκτυπο στον ε, προπολογισμό. Υπάρχουν βέβαια μακροχρόνιες προεκτάσεις που θα γίνουν εμφανείς μέσα σε δεκαετίες. Πράγματι, οι οργανισμοί συμβάλλουν ε, στο βαθμό που του αναλογεί ε, στα, στα εξωτικά ταμεία, αλλά από πλευρούς, πλευράς ε, εποπτείας δεν θα πρέπει αυτό να το παραμελήσουμε. Τώρα, για τον καθορισμό των τελών, κατά πόσο δηλαδή τα τέλη αυτά ε, αντανακλούν και το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στην αγορά, νομίζω ότι αυτό είναι... Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι η ευθύνη της ότι υπάρχει τέτοια ευθύνη της εποπτείας. Σίγουρα θα αναφερθεί και από τους επόμενους ομιλητές. Έχουμε ε, στους ε, πλήρους αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς και την δημιουργία αποθεματικών που νομίζω ότι είναι εδώ ευθύνη γενικής εποπτείας των θεσμικών οργάνων. Θα μείνω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρέσα ε, για αυτήν την ε, πρώτη γενική εικόνα. Άκουσα επίσης ότι εκπροσωπείται εδώ και το ελεγκτικό συνέδριο και χαίρομαι ιδιαίτερος που παρευρίσκεται εδώ. Και δεύτερος ο κύριος Σπανιόλη από την Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων. ΕΦΣΑ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ε, με χαρά συμμετέχει σε αυτή την ε, συνεδρίαση. Ε, προεδρεύουμε στο δίκτυο των αποκεντρωμένων οργανισμών για φέτος και φυσικά μας ενδιαφέρουν τα θέματα τα οποία συζητούνται εδώ σήμερα. Παρά το γεγονός, αν θέλετε δώστε μου το τηλεκοντρόλ για τις διαφάνειες. Um, this workshop uh, Το εργαστήριο αυτό εξετάζει κυρίως ε, υπηρεσίες και οργανισμούς που χρηματοδοτούνται μέσω αμοιβών. Ε, είναι 45 οι υπηρεσίες στο σύνολο και μόνο πολύ μικρό ποσοστό χρηματοδοτείται μέσω αμοιβών. Ε, όσον αφορά το ποσοστά, όπως βλέπετε και από τις διαφάνειες, το 38% του προσωπικού όμως των υπηρεσιών πληρώνονται μέσω αυτών των αμοιβών. Ε, αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για το δίκτυο συνολικά και είναι επίσης πολύ σημαντικό και για το δίκτυο διότι πέραν των θεμάτων που συνδέονται άμεσα με την διαχείριση αυτών των αμοιβών, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες πρέπει να ασχοληθούν και με άλλα θέματα διαχείρισης σπόρων που αφορούν και όλους τους υπόλοιπου οργανισμούς. Και φυσικά έχουμε κοινέ προκλήσεις στον τομέα αυτό και θα πρέπει να πω ότι όπως υπενθύμησαν και οι προλαλήσαντε, το θέμα των αμοιβών και τα θέματα των εναλλακτικών πηγών ε, χρηματοδότησης είναι ένα θέμα το οποίο στο μέλλον ε, θα αφορά όλο ένα και περισσότερους οργανισμούς και υπηρεσίες ε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο και ω δίκτυο βεβαίω είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να εξετάσουμε και να δούμε φυσικά και να συζητήσουμε με τα μέλη μας πώς μπορούμε να έχουμε πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα ενταχθούν στο σύστημα στο μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η όλη συζήτηση για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται μέσω αμοιβών και τα όσα είπε και ο προλαλής σας ε, αφορούν κυρίως την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εποπτείας, πώς θα εφαρμόζονται οι κανόνες και επίσης πώς θα έχουν και ταυτόχρονα οι οργανισμοί την ευελιξία να διαχειρίζονται καταλήλως τις δραστηριότητές τους. Και αυτό φυσικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται μέσω αμοιβών, αλλά και για τους υπόλοιπους οργανισμούς. Οι συζητήσεις αυτές λοιπόν στον κόσμο της χρηματοδότησης μέσω αμοιβών ουσιαστικά δίνουν και κάποιες απαντήσεις οι οποίες θα μπορούσαν σε κάποιες περιπτώσεις να επεκταθούν και σε άλλους οργανισμούς. Η παρουσίασή μου θα είναι από το υψηλότερο επίπεδο, επίπεδο δικτύου δηλαδή. Προσπαθούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα για τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν και ε, να δώσουμε και κάποιες υποδείξεις για το πώς ε, ε, βλέπουμε να εξελίσσεται το μέλλον, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών αυτών. Αν δείτε τι έχει συμβεί από το 2012 και μετά, Ξεκινούμε με ε, σημείο κίνηση το 2012, διότι είναι ίσως καλή χρονιά, είχαμε την κοινή προσόγγιση, τον χάρτη πορείας και ήρθε και μετά από τη σύσταση των πιο πρόσφατων οργανισμών, επομένως ε, σταθεροποιήθηκαν και λίγο τα αριθμητικά στοιχεία. Την τελευταία πενταετία λοιπόν, ε, ο τρόπος με τον οποίο καθορίζαμε πώς γινόταν η διαχείριση και η χρηματοδότηση των οργανισμών ήταν ε, καταρχά η κοινή προσέγγιση και η όλη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, τις περικοπές στο προσωπικό, ε, το πάγωμα του προπολογισμού και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 που μόλις αναφέρθηκε. Mm-hmm. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν ουσιαστικά ε, αποτέλεσαν και το ε, μοχλό κίνησης των δραστηριοτήτων. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, σίγουρα πρόκειται για επιτυχημένη ε, ιστορία. Το 99,7% των δράσεων που ξεκίνησαν ή εφαρμόστηκαν έχουν σχεδόν περατωθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από πλευρά δικτύου. Αυξήθηκε η διαφάνεια και η λογοδεσία και η συνοχή των οργανισμών. Επίσης, ε, συντονισμός και συνεργασία. Ε, αυτά αυξήθηκαν πάρα πολύ σημαντικό και, αυτό είναι σίγουρα θετικό. Όσον αφορά τα αρνητικά, αν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε έτσι, υπήρχε αύξηση του γραφειοκρατικού άχθους, κάτι το οποίο επεσήμανε ούτως ή άλλως ε, το δίκτυο. Επίσης, άλλαξαν και κάποιες επιβαρύνσεις στο συντονισμό, το, το οποίο και πάλι βάρινε το δίκτυο. Και επίσης, πρέπει να πω ότι Υπάρχει πρόσφατη έκθεση της απαλλογής του 2015, η οριζόντια έκθεση ε, για τους οργανισμούς ε, αναγνώρισε ότι πρέπει να αυξηθεί το, το προσωπικό για το συντονισμό, η γραμματεία δηλαδή, να έχουμε περισσότερο προσωπικό ώστε να διασφαλίσουμε ότι το δίκτυο θα μπορεί να απαντήσει σε όλα τα αιτήματα που έρχονται από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για το συντονισμό του έργου των ε, οργανισμών και των υπηρεσιών. Υπήρχε επίση και έλλειψη ευελιξία, ήταν περίπλοκα τα πράγματα, κυρίως για τον κανονισμό ε, των υπαλλήλων και τον δημοσιονομικό κανονισμό. Μετατοπίστηκαν κάποια ε, ε, δαπάνες, κυρίως για τις εξωτερικές αξιολογίες και ελέγχους. Και επίσης υπήρχαν και τα θέματα κοινή συμμόρφωσης, μεταφορές από προηγούμενα έτη κλπ. Αν δούμε το επόμενο στοιχείο, το οποίο ήταν βασικό για τις δράσεις του δικτύου την τελευταία πενταετία, το θέμα των περικοπών του προσωπικού με την προσέγγιση ε, ε, η οποία θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι κοινή και εδώ το αποτέλεσμα είναι ε, θετικό. Οι υπηρεσίες έχουν υπερβεί το 5% και έχουν φτάσει πολύ κοντά και στο 10% από ό,τι αποδεικνύεται στις περικοπές προσωπικού παρά το γεγονός ότι εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτή το, ε, την δυνατότητα να ε, μεταφέρετε και να αποσπάτε προσωπικού αλλού. Ε, η μείωση του προσωπικού ούτως ή άλλως έχει πάει όσο θα έπρεπε. Είμαστε πολύ, καλά, πολύ κοντά στο 10% και υπήρξαν και κάποια θετικά αποτελέσματα από την όλη αυτή διαδικασία γιατί πιέστηκαν οι οργανισμοί για αυξημένη αποτελεσματικότητα και συνεργασία και ενισχύθηκε η προσέγγιση αυτή ε, one size fits all. Ε, επομένως βλέπουμε μέχρι ποιο σημείο έχουμε φτάσει και πόσο μεγάλη πρόοδο έχουν επιτελέσει οι οργανισμοί στη ε, διαχείριση των οργανισμών. Τώρα, όσον αφορά τα αρνητικά, επειδή ακριβώς ακολουθήθηκε νέα προσέγγιση, βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες αρνητικές προτεραιότητες, πολύ συχνά ε, δεν οδηγούσαν στις κατάλληλες κατευθύνσεις από πλευράς πολιτικής. Ήταν μάλλον τακτική η προσέγγιση και όχι στρατηγική για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και ε, φυσικά κάτι που είναι πολύ σημαντικό υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξωτερικής ανάθεσης και επισφαλούς εργασίας. Ε, κάποιες απαραίτητες θέσεις αντικαταστάθηκαν από συμβούλους, από προσωρινό προσωπικό, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη. Ε, βλέπετε επίσης και στην τελευταία ε, παύλα ότι υπάρχουν και κάποιες πολλωμένες θέσεις οι οποίες προέκυψαν στη συζήτηση περί υπολογισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα το οποίο εμείς δεν θεωρούμε ότι ε, είναι αραγός της συνεργασίας ως δίκτυο και θεωρούμε ότι θα έπρεπε ίσως να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε διαφορετικό κλίμα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, Ας δούμε λίγο πώς ε, θα θέλαμε να εξελιχθεί υπό ιδανικές συνθήκες η κατάσταση στο μέλλον. Έχουμε ένα όραμα και έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι έχουν σχέση με το όλο θέμα και θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ε, το μοχλό καθοδήγηση στο μέλλον. Τα αναφέρουμε εδώ, μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα. Ε, κοινέ υπηρεσίε και δυνατότητες. Ε, αυτή τη στιγμή είναι κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη προτεραιότητα του δικτύου και των οργανισμών και των υπηρεσιών. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και υπάρχουν και άλλα πράγματα στα σκαριά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κατάλογος υπηρεσιών και δυνατοτήτων που ε, είναι κοινέ μεταξύ των οργανισμών και είναι πολύ εκτεταμένη αυτή η διαδικασία επιμερισμού τις χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες. Έχουμε κάποια ε, ενδιαφέροντα παραδείγματα για χρήση πόρων από αυτό το αποθεματικό. Ε, για παράδειγμα, ε, απάντηση σε καταστροφές. Έχουμε και δημόσιους διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν έρθει από έναν επιτυχή διαγωνισμό που κάναμε πέρσι για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε πολύ ουσιαστική αποταμίευση πόρων. Και το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, αλλά θέλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί νομίζω ότι ε, μπορούμε να έχουμε πολλά ωφέλη με τη συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που είναι μικροί, ευέλικτοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο καινοτόμους ε, τρόπους εξωτερικής ανάθεσης, μπορούν να εξετάσουν άλλους ε, τρόπους συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι λίγο πιο βραδικίνητη γιατί φυσικά είναι πιο μεγάλος οργανισμός αλλά έχει και την κρίσιμη μάζα. Όταν γίνονται λοιπόν πράγματα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αντίκτυπος ε, για την αποτεμίευση και την αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Επίση πρέπει να πω ότι εξετάζουμε πολλού νέου τομεί συνεργασία και ανταλλαγή υπηρεσιών με του άλλου οργανισμού και υπηρεσίε, Ξεκίνησαν με θέματα όπω είναι η πληροφορική και οι πόροι όπου μπορούμε να έχουμε κάποιες κοινέ υπηρεσίες, αλλά θέλουμε να τα επεκτείνουμε και στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων να γίνεται διαχείριση από κοινού, κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα και επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες βασικές δραστηριότητες από κοινού. Παραδείγματο χάρη, εμείς ως ΕΦΣΑ ασχολούμαστε με την επιστήμη και συνεργαζόμαστε και με τους άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με επιστημονικά θέματα, διότι θέλουμε και εμείς να ε, έχουμε συνεργασία. Γίνεται ανταλλαγή εμπειρογνωμένων, υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες και αυτά φυσικά είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα θέλαμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Εάν ε, δείτε τον άλλο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε ως δίκτυο, κυρίως ε, εστιάζουμε στην απόδοση. Θέλουμε να έχουμε ε, διαχείριση που θα βασίζεται σε αποτελέσματα, προπολογισμό που θα βασίζεται στα αποτελέσματα. Αυτό προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ θεωρώ ότι εκφύσεω οι υπηρεσίε και οι οργανισμοί, επειδή είναι μικροί, πιο ευέλικτοι και έχουν και τη δυνατότητα να ε, διαχειριστούν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, ε, μπορούμε να κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Φέτος ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα μοντέλο ορίμανσης μέσω του οποίου όλοι οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες θα μπορούν να δουν τι δυνατότητες χρειάζονται και τι συνέπειες έχει αυτό, αν δηλαδή περάσουν από τη διαχείριση του προπολογισμού που βασίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και σε συνεισφορές, ε, σε διαχείριση προπολογισμού που θα επικεντρώνεται σε αποτελέσματα ε, και φυσικά σε αντίκτυπο. Αυτό ε, σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες, να δούμε κάποιους βασικούς δείκτες απόδυσης οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και επίσης να δούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά είναι στα σκαριά, είναι εν εξελίξη και με χαρά διαπιστώνουμε ότι συμμετέχουν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα στις δραστηριότητες που κάνουμε εμείς ως δίκτυο. Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε εδώ ότι ε, σίγουρα είμαστε και προετοιμασμένοι να ξεκινήσουμε ένα ε, πιλωτικό πρόγραμμα ε, προϋπολογισμού βάση απόδοσης ε, και ξέρουμε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο σε θεσμικό επίπεδο. Όλα αυτά βεβαίως ε, στόχο έχουν να ε, ε, έχουμε αλλαγή στην προσέγγιση και να μην μετράμε πόσο προσωπικό έχουμε, αλλά να έχουμε μακροπρόθεσμη διαχείριση. Οι περικοπές στο προσωπικό κατέδειξαν ότι το να βασιζόμαστε στο πόσους υπαλλήλου έχουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο και φυσικά είναι και πολύ αυστηρή η όρη και δεν μας εξυπηρετεί. Εδώ έχουμε την πτυχή της χρηματοδότησης μέσω αμοιβών. Δεν θα ε, πω περισσότερο. Είναι οι συνάδελφοι από την ΕΑΣΑ και τη ΣΥΠΙΟ που θα σας πούν περισσότερα. Αλλά και πάλι εδώ ε, θα έπρεπε να πω ότι κυρίως ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να επεκτείνουμε την όλη συζήτηση για άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Υπάρχουν ε, κάποιοι οργανισμοί. Εμείς ως δίκτυο δεν έχουμε σαφή θέση, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να τα εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ένα άλλο τμήμα του οράματος που έχουμε για το μέλλον είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και σαφέστατα στην πρώτη έκθεση για την απαλλαγή του 2015 που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχει τομεακή θεματική προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε κάποιες ομάδες οργανισμών υπηρεσιών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, που συνεργάζονται ε, και φυσικά Είναι και λογικό να διαχειριζόμαστε και τους πόρους ε, με αυτόν τον τρόπο, βάση δηλαδή θεματικής τομεακής προσέγγισης. Να εξετάζουν δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν αυτοί οι οργανισμοί από κοινού και φυσικά ε, τους ευρύτερους τομείς πολιτικής και αυτή η τομεακή θεματική προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμαστεί τρόπον την Α, κατά την εκτέλεση του προπολογισμού, κατά την εξέταση της απόδοσης και φυσικά την απαλλαγή. Είναι πολύ ε, περίπλοκος ο τομέας, αλλά θα θέλαμε να κάνουμε συζητήσεις, να δούμε αν μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό το θέμα. Τώρα, ε, απλούστεροι και πιο ευέλικτοι ε, δημοσιονομικοί κανονισμοί για κανονισμοί προσωπικού. Αυτό το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει ότι ορισμένες φορές υπάρχουν πάρα πολλές αγκυλώσεις που ε, καθυστερούν την όλη διαδικασία, αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συζήτηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού και ελπίζουμε ότι πολλά από τα θέματα που εξετάζουμε και εδώ θα μπορούσαν να επιληθούν. Στον κανονισμό του των υπαλλήλων ε, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αναθεώρηση. Αλλά όσον αφορά τους εκτελεστικούς και τους ε, ε κανόνες, ε, θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες και να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ίσως στους κανόνες. Όλα αυτά νομίζω αποδεικνύουν ότι κινούμαστε ως ε, το ιδανικό κλίμα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων και φυσικά ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα επιτρέψει να έχουμε κοινό λεξιλόγιο και να έχουμε διάφανο διάλογο, να εξετάσουμε τα θέματα προπολογισμού και να δεσμευόμαστε όλοι από κοινού και να θεωρούν όλοι ότι το δίκτυο είναι ένα έμπιστο εταίρος που μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό τη κατανομή του προπολογισμού ε, και να μπορούμε να τα αποφασίσουμε αυτά σε κλίμα πλήρου συνεργασία, να μοιήσουμε τακτικέ κινήσει και να επικεντρωθούμε σε στρατηγικό επίπεδο βεβαίως. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν με αυτή την επιθυμία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Vielen herzlichen Dank. Ευχαριστούμε πολύ ε, για αυτήν την ε, παρουσίαση αλλά και για τα οράματα τα οποία ε, υπάρχουν και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια που είναι η καθηγήτρια Έλεν Βος η οποία είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος για ΤΑΡΝ Έχετε το λόγο. Thank you. Well, that's... Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα όρο ο οποίο χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία για μια διαδικασία όπου ε, η εκτελιστική ε, εξουσία δίνεται στου οργανισμού για να μπορέσουν να επιτελούν εκτελιστικά έργα. Ε, είναι ένα γνωστό λοιπόν όρο στην λογοτεχνία και πιστεύω ότι σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλο αυτό έχει γίνει χαρακτηριστικό ε, της ε, εκτελεστικής της Ένωσης ε, το πρόγραμμά μας, το TARN, εξετάζει όλη αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα να σας ε, ε, πω, ε, να σας εξηγήσω το τι ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο ε, δίκτυο ακαδημικής έρευνας που μελετά τις υπηρεσίες αυτές και θα ήθελα να σας μιλήσω επίσης για τη διαδικασία της απαλλαγής ως ένα εργαλείο για τις υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από αμοιβέ. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Ζαμονέ ε, Είναι ένα ερευνητικό δίκτυο, ε, ένα δίκτυο πληροφόρηση ε, το οποίο λειτουργεί στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα διεθνικό επίπεδο. Αποτελείται από εννέα ακαδημαϊκού εταίρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φέρει ε, ακαδημαϊκούς ε, νέους αλλά και γνωστούς οι οποίοι ασχολούνται με, με την πληροφόρηση, με την νομοθεσία. Το Τάρν λοιπόν έχει μια διτή αποστολή από την μία προωθεί ε, τις ε, διαλειτουργικές ε, αποστολές των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας να ενσωματώσει τις λειτουργικές προσεγγίσεις για να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ του ακοδημαϊκού αλλά και αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν την όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν το ΤΑΡΝ δεσμεύεται να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών, ε, των νομοθετών, ε, τη κοινωνία των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μέρη για την ανταλλαγή απόψεων ε, προσφέρει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών σε στρογγυλές τράπεζες. Επικεντρώνεται σε τέσσερα θέματα αφενός επικεντρώνεται στην, στον καθορισμό ε, της ε, υπεροποίησης ε, της εκτελεστικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπρόσθετα αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες ως μεσολαβητές των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της. Ε, αφορά επίσης την συνταγματικότητα, τις ε, εξουσίες και την νομικότητα ε, των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζουμε δηλαδή ποιο είναι το συνταγματικό τους πλαίσιο και θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί καλύτερα στις συνθήκες. Επίσης έχουμε αναπτύξαμε τον, έναν κανόνα ο οποίος ορίζει τη λειτουργία τους και αντιμετωπίζει επίσης ζητήματα τα οποία αφορούν τη διάβγεια και την ε, λογοδεσία. Επίσης επικεντρωνόμαστε στην ε, διεθνή διάσταση της δραστηριότητας των υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ έχουμε ε, την έρευνα στην οποία επικεντρώνεται το ΤΑΡΝ σχετικά με την νομική τους βάση σχετικά με τις δραστηριότητες που κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τους ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο και τέταρτον ζούμε, ε, την ε, λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών ε, γύρεται ένα κοινό ερώτημα το πώς μπορούν να οργανωθούν καλύτερα ούτως ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητα επεκτείνεται πέρα από, την, από τις τεχνικές δυνατότητες για να περιλάβει ταυτόχρονα και εσωτερικά ζητήματα όπως είναι η αποτελεσματικότητα του προπολογισμού, ζητήματα κατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών παραγόντων καθώ επίσης και διαχείριση προσωπικών προσωπικού αλλά και την ορθή διαχείριση. Επίσης εκδίδει ε, έντυπα, ε, οργανώνει ε, συνέδρια, συμμετέχει σε blog, συγκεντρώνει, διοργανώνει συναντήσεις ακαδημαϊκών για να συζητήσουν πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Τα μαθήματα αυτά οργανώνονται από τους εταίρους του ΤΑΡΝ στο Όσλο, στο Παρίσι, τη Ρώμη, το Βερολίνο ε, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης μια βάση δεδομένων ε, για τη βιβλιογραφία αλλά και ε, τα και νέα σχετικά με το έργο της υπηρεσίας. Έχοντας λοιπόν εξηγήσει την αποστολή και τις δραστηριότητες της ΣΤΑΡΝ και χαίρομαι ιδιαίτερος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Θα ήθελα επίσης τώρα να στραφώ στο ζήτημα της δημοκρατικής λογοδοσίας των υπηρεσιών της Ένωσης και ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της απαλλαγής ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε ε, ε, στο ζήτημα της κοινή προσόγησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καταλήξει στο ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καλύτερα ε, να σκεφτούμε καλύτερα μηχανισμούς λογοδεσίας. Ακαδημαϊκοί λοιπόν έχουν παρατηρήσει ότι ε, υπάρχει ένα κενό λογοδοσία πάνω σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο θα θέλουμε να το διαχωρίσουμε στην πολιτική λογοδοσία, τη διοικητική λογοδοσία, την οικονομική λογοδοσία, καθώ επίση και την νομική λογοδοσία. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε γι' αυτό λεπτομερέστερα στη συνέχεια. Αναμφίβολα το Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο στη διασφάλιση της εποπτείας ε, των υπηρεσιών της Ένωσης στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο της απαλλαγής ε, για να τονίσει ένα προβληματικό ζήτημα όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς η ανεξαρτησία του προσωπικού ε, και ε, του προσωπικού. Η χρήση αυτού του εργαλείου από το Κοινοβούλιο έχει οδηγήσει οργανισμούς όπως η ΕΦΣΑ να αντιμετωπίσουν και να απτύξουν μια, πολιτική η οποία βασίζεται στην ανεξαρτησία όταν αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων για παράδειγμα. λαμβάνοντας υπόψη μας ε, την ε, ενημέρωση αυτών των ε, υπηρεσιών είναι σημαντικό να να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τους οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε εργαλεία εποπτείας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό η δέσμευση για την διαφάνεια ε, καθώς επίσης και η ανάγκη να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στις λήψεις αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εργαλείο της απαλλαγής θα είναι ένα πολύ καλό μέσο εποπτέως το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε, όλες τις, ε, σε όλους τους οργανισμούς ε, της Ένωσης καθότι είναι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση και άλλων ε, μηχανισμών εποπτείας. Ε, το ΤΑΝ κατάληξε ότι θα πρέπει να υπάρξει περιττέρω ε, έρευνα σχετικά με τη λογοδεσία αλλά και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουμε το 2018 στο ΤΑΝ. Επίσης μπορούμε να προσφέρουμε μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των εργαζομένων αλλά και των ακαδημαϊκών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βόσ για την εικόνα την οποία μας δώσατε ε, Βάσει της τελευταίας ε, σας πρότασης θεωρώ ότι οι οργανισμοί ε, που χρηματοδοτούνται μερικώς αλλά και πλήρως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία. Δεν θα πρέπει να το θεωρούμε όλο αυτό αυτονόητο επειδή χρηματοδοτούνται από αμοιβέ και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο συμφωνούμε όλοι στο Κοινοβούλιο και ακολουθεί ο κύριος Μάρτιν Εκβάτο ο οποίος είναι επικεφαλής του Κοινοτικού Γραφείου Φοιτικών ποικιλιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της σημερινή εκδήλωσης και για την πρόσκληση που απευθύνω στο πρόσωπό μου. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους ευρωβουλευτές ε, να συνομιλήσουν με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και συγκεκριμένα σε αυτούς που βασίζονται ε, σε αμοιβέ. Εμείς είμαστε πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός ε, και ε, παραδοσιακά είχαμε πολύ περιορισμένες επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως εφόσον το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει ε, τον προπολογισμό ε, του Κοινοτικού Γραφείου Φοιτικών Ποικιλιών και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία απαλλαγή. Όμως, μετά την υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο εμπλέκεται σε όλα τα νομοθετικά ζητήματα και για το κοινοτικό μας γραφείο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Ακούσαμε τις ε, γενικότερες ε, επιφυλάξεις και προβληματισμούς που ανέφεραν ε, οι επικεφαλής των οργανισμών που έλαβαν τον χώρο, το λόγο προηγουμένως. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι να μιλήσω λίγο για, για αυτές τις μερικώς ή πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες, αλλά να μιλήσω και για τις προκλήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ενός ε, δυναμικού ε, αυτοχρηματοδοτούμενου οργανισμού. Θα διατρέξω αυτά τα ζητήματα συντομία, στο χρόνο που μου απομένει, παρότι είναι αρκετά. Επομένω, ε, η δική μας οπτική γωνία, η απαλλαγή, διαχείριση αποθεματικών, ανθρώπινη πόρη, τεχνικά ζητήματα ε, και τα βασικά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, με περηφάνεια μπορώ να πω ότι εμεί χειριζόμαστε το μεγαλύτερο σύστημα φοιτικών ποικιλιών στον κόσμο. Είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, όπω ανέφερα. Και με αυτό εννοώ ότι όχι μόνο δεν λαμβάνουμε πόρους από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά όπως ε, επισήμανε και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλουμε στα στοιχειωτικά ταμεία και έχουμε και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ε, εισφορές. Από έναν προπολογισμό 80 εκατομμυρίων, το 1,6 εκατομμύριο ε, καταβάλλεται για, στα συνταξιδοτικά ταμεία. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα στο μέλλον. Για να σας δώσω μία γενική εικόνα, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε λάβει 60.000 αιτήσει. 26.000 ενεργούς ε, τίτλους έχουμε, κάθε χρόνο περίπου 3.500 ε, αιτήσει. Καταβάλουμε, μάλλον στέλνουμε, κόβουμε τιμολόγια ε, στις τάξεις των 40.000 ε, κάθε χρόνο και έχουμε έναν και έχουμε μόνο 45 ε, υπαλλήλου, παρότι είναι σκληρά εργαζόμενοι. Μερικέ φορέ υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο ο κατάλληλο τρόπο εφαρμογή ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι μέσω ενό ευρωπαϊκού οργανισμού. Εμεί θεωρούμε ότι όντω έτσι είναι. Ε, μπορούμε πολύ γρήγορα να ανταποκριθούμε στι ανάγκε των πελατών μα Έχουμε εξαιρετικά ικανούς ε, υπαλλήλους, έχουμε ε, και χαίρουμε μεγάλου σεβασμού στον ε, κλάδο μας και οι ετούντε μπορούν πολύ πιο εύκολα, αντί να κάνουν 28 διαφορετικές αιτήσει σε, όλες τις, σε όλα τα κρατημέλη, κάνουν μία αίτηση σε μία γλώσσα με μία διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο. συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη γιατί η τεχνική εξέταση είναι στο δικό μας σύστημα. Θεωρούμε ότι αυτό το κάνουμε για μία αμοιβή που είναι εύλογη. Δύο λόγια τώρα για την διακυβέρνηση και την απαλλαγή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ισχυρή εποπτεία για όλου του ευρωπαϊκού οργανισμού. Είμαι πεπισμένο ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων. Ε, Όμω και η χρηστή ε, δημοσιονομική διαχείριση θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη σημασία για οργανισμού όπω ο δικό μα. Δεν πρέπει απλώ να ακολουθούμε τον δημοσιονομικό κανονισμό, που βεβαίω και πρέπει να κάνουμε, αλλά θα πρέπει ξεκάθαρα να λέμε και στους πελάτες μας ότι ε, εμείς εφαρμόζουμε τους, ε, τις αρχές ε, της χρηστής διαχείρισης στις καθημερινές μας λειτουργίες. Και έχουμε μάλιστα και την απαλλαγή από το Διοικητικό Συμβούλιο στο κοινωνικό μας γραφείο και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευρύτερη διαδικασία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω υπερασπίζεται ε, τα δικαιώματα ε, των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τις, ε, και τις απαλλαγές, όμως σε μια μικρότερη κλίμακα η παρουσία του κλαδού που χρηματοδοτεί το CPVO για την έγκριση του προπολογισμού και για την απαλλαγή σε τη αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, όχι μόνο είναι δικαιολογημένη, θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για άλλου οργανισμού. Δεν ξέρω αν εδώ σα προκαλώ. Όμω η απαλλαγή γίνεται βάσει εκθέσεων του Λεκτικού Συνεδρίου και να υπερθυμίσω ότι ε, μάλιστα περνούν ε, τον ίδιο χρόνο στο δικό μας γραφείο που είναι μικρό σε σχέση με ε, τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Όμω με τα χαρά θα θέλουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εποπτεία και την ενημέρωση. Όμω δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία τη ε, συμπερίληψη και, ε, και όσων συνεισφέρουν οικονομικά σε αυτή τη διαδικασία που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν ε, με μεγάλη προσοχή πώ δαπανώνται τα χρήματα. Μεταξύ άλλων και μέσω του αριθμού των υπαλλήλων. Βέβαια, όταν πληρώνει για κάτι, θε να ξέρει τι συμβαίνει. Να έχει εικόνα τη κατάσταση και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό συμβαίνει γενικά και όσοι μας χρηματοδοτούν αλλά και τα κρατη με μεγάλη προσοχή εξετάζουν τα όσα κάνουμε. Εμείς έχουμε πάντα ως στόχο έναν ισοσχελισμένο προπολογισμό. Όμως πάντα, έτσι συμβαίνει με, τις, ε, με τους οργανισμούς ε, που βασίζονται στην αγορά, πρέπει να ισοσχελίσουμε τον προπολογισμό μεσοπρόθεσμα και όχι σε αιτήσια βάση. Από αυτήν την άποψη λοιπόν ε, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός αποθεματικού. Ε, είναι λοιπόν ένα εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε, μία, ε, έχουμε κάποιες ταμιακές ροές ε, κατά περιόδους που είναι λιγότερες αμοιβέ από τις αναμενόμενες και όταν έχουμε απαραίτητα προγράμματα υποδομών ή αναπτυξιακά προγράμματα. έχουμε ένα σχετικά ευέλικτο σύστημα διαμόρφωσης των αμοιβών βάσει του δικού μα Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την επεξεργασία των τροποποιήσεων και αυτό έχει επιτρέψει στο γραφείο μας τα τελευταία χρόνια από ένα παθαματικό 12 εκατομμύριων ευρώ να περάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ. στις 500.000 ευρώ. Ε, και ε, αυτό βλέπετε ότι έχουμε αυξήσει τώρα τις αμοιβέ. Και έτσι φτάνουμε σε μια κρίσιμη κατάσταση ό,τι αφορά το ποσό του αποθεματικού. Δεν ε, λειτουργούμε ως τράπεζα λοιπόν για τους πελάτες μας. Επανέρχομαι τώρα στο πιο σημαντικό για μένα ζήτημα για τον οργανισμό μας. Το δίκτυο οργανισμών, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, συμφώνησε για τον στόχο το 5%, συν ένα επιπρόσθετο 5% ε, για την ανακατανομή του προσωπικού, το οποίο για λόγους που ξέρετε έχει τύχει κάποιας ε, διαφωνίας. Όμως για τους πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς αυτό το επιπρόσθετο 5% είναι ακόμα πιο παράλογο, γιατί εμείς δεν μπορούμε νόμιμα να καταβάλουμε χρήματα προ τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και δεν γίνεται να λαμβάνουμε λιγότερα χρήματα από τον προπολογισμό. Αν κάνουμε περικοπέ του 10, 20, 30% και του 90% του προσωπικού, αυτό δεν επηρεάζει ε, κατά οποιονδήποτε τρόπο τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Γιατί πώ μπορώ λοιπόν να εξηγήσω στο προσωπικό μου ότι πρέπει να κάνουμε περικοπέ 5% και να του πω ότι είναι ε, ο μηχανισμό ε, ανακατανομή, στον οποίο δεν μπορούμε εμεί κάπω να συμβάλλουμε. Αυτό είναι λοιπόν μια αντίφαση. Είναι διαφορετική λοιπόν η δομή, οπότε και η ανάλυση θα πρέπει να είναι διαφορετική για να βασίζεται στην πραγματική κατάσταση. Μπορείτε να πείτε ότι ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση ε, ενό οργανισμού θα πρέπει να υπάρχουν περικοπέ του προσωπικού για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα που τελικά ε, θα γλιτώσει υψηλέ αμοιβέ ε, για την βιομηχανία, για τον κλάδο. Εντάξει, σωστή προσέγγιση. Όμω αυτό με την προπόθεση ότι υπάρχει ένα status quo που δεν υπάρχει όμω εμείς ε, στο δικό μας κλάδο έχουμε αυξήσει την ε, ζήτηση. Οι πελάτες μας ε, αποτελούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από πολυεθνικές. Όμως το κοινό σημείο που έχουν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερα στους επιβίω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όμως στην τελευταία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου μας προτείναμε να μην υπερβούμε το 5% αυτή την περικοπή που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει και ο κλάδος συμφώνησε. Θεώρησε ότι όντω θα πρέπει να έχουμε αυτούς τους ανθρώπινους πόρους. Επομένω, έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Αυτοί που χρηματοδοτούν τους επιβιώσεις συμφωνούν ε, για το πάγωμα ε, των ανθρωπινών πόρων, αλλά μας είπαν από την Γενική Διεύθυνση Υπερβολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι παράλογο και είναι ένα κακό παράδειγμα διαχείρισης για να σας δώσω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Τα κράτη-μέλη απαιτούν περισσότερα αποτελέσματα από τον Frontex. Είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν ε, ε, τέτοια αποτελέσματα, επομένω δίνουν περισσότερου πόρου. Λογικό. Ο κλάδο απαιτεί περισσότερα αποτελέσματα από τον CPVO. Είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το τίμημα για να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, αλλά ε, δεν καλύπτεται αυτό από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό δεν είναι λογικό. Επομένω, σας χαιρετίζω για την ε, ε, πρωτοβουλία για το πιλωτικό έργο για τον ΙΑΖΑ, γιατί έτσι ταυτοποιούμε τους πραγματικές, τις πραγματικές ανάγκες με συναφείς δείκτες και μπορούμε να συζητήσουμε το μοντέλο που θα ακολουθηθεί, όμως ε, η αρχή της διασύνδεσης των πόρων με τις πραγματικές, ε, ε, την πραγματική ζήτηση είναι, πιστεύω, αυτονόητο. Δεν πρέπει να περιμένουμε όμω για τα τελικά αποτελέσματα του πολιτικού έργου. Πρέπει να γίνει αυτό άμεσα γιατί χρειαζόμαστε τώρα αυτού του πόρου. Δυο λόγια τώρα για το φόρτο εργασία πριν ολοκληρώσω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στην οθόνη, αλλά το έχετε και στο υλικό που σας έχουμε διαβιβάσει. Οι βασικοί δείκτες ε, φόρτου εργασίας για το CPVO είναι εδώ, που επηρεάζουν ε, άμεσα και τις ανάγκες μας ανθρώπινο δυναμικό. Και βλέπετε εδώ το σχεδιασμό που έχει ε, πέσει. Επομένω, η κατάσταση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό έχει σταθεροποιηθεί ή ακόμα και έχει πέσει, παρά το γεγονό ότι έχουμε 40 ώρες εργάσιμου χρόνου που δεν ε, καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Είμαστε λοιπόν ένας μικρός οργανισμός ε, που καλύπτουμε τις ανάγκες της βιομηχανίας, όμως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τους ίδιους ε, διοικητικούς στόχους ή τους ίδιους περιορισμούς με μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Χρειάζεται όμω ε, μια κρίσιμη μάζα για να ε, λειτουργήσει ένα τέτοιο οργανισμό. Και εδώ είναι πραγματικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, στο CPVO μιλούμε μόνο για ε, περικοπή δύο-τριών θέσεων και μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι εύκολο. Όμως, κάθε υπάλληλο μας είναι πολύ σημαντικός για μας. Και θα ήθελα να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν υπό αυτό το πρίσμα την κατάσταση. να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με την ανακοίνωση του 2013. Θεωρώ ότι είναι παράλογο παρά το γεγονό ότι εμεί ε, δείχνουμε ότι λειτουργούμε πολύ καλά και έχουμε και τη στήριξη του κλάδου. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, να μην πω λοιπόν στα υπόλοιπα ζητήματα που ε, έχω συμπεριλάβει στην παρουσίαση για ε, υπό τον δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε το δικαίωμα να έχουμε παθηματικό, αλλά προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Τέλος, ορισμένα κύρια μηνύματα. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερω ε, το πιλωτικό πρόγραμμα για τον ΙΑΖΑ, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, πρέπει να βρούμε το σωστό επίπεδο ελέγχου με έναν ισορροπημένο τρόπο και πρέπει να επικεντρωθούμε στην χρηστή δημοσιονομική ε, διαχείριση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή σας ε, παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε κι εσείς να έχετε το μοντέλο σαν την, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας. Δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Τα κράτη-μέλη δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένα στην αρχή, αλλά τελικά βρήκαμε μια σωστή λύση. Τώρα έχουμε τον κύριο Ζαν Μισελ Μαστιού από την ε, ΕΑΣΑ. Είναι αναπληρωτής διευθυντής πόρων και υποστήριξης, επικεφαλής των του τμήματο ε, χρηματοοικονομικών και προμηθειών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια τη Αεροπορία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι προσκαλέσατε τον ΕΑΣΑ και ε, μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τι κάνουμε και πώς μπορούμε να δούμε τις ε, διάφορες ε, δημοσιονομικές πτυχές. Πριν ε, αναφερθώ λοιπόν στα χρηματοοικονομικά και στη διακυβέρνηση, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία εικόνα του τι ακριβώς κάνει η ΆΣΑ. Εκ πρώτη βλέπετε ότι δραστηριοποιούμεθα για πάνω από 15 χρόνια. Ε, έχουμε δράσει στην Κολονία, στη Γερμανία, Έχουμε την έδρα μας εκεί, έχουμε και κάποια γραφεία ε, ανά τον κόσμο, στις Βρυξέλλες, στη Washington, στο Μόντρεαλ, έχουμε και γραφείο στη Σιγκαπούρη. 800 άτομα απασχολούμε ε, στην κολονία. Οι περισσότεροι είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα αεροπορίας και στα συστήματά μας ε, περιλαμβάνονται 32 κράτη-μέλη, 28 ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 επιπλέον που συνεισφέρουν και αυτά στον οργανισμό. Η αποστολή του οργανισμού είναι Βεβαίω και όλοι ενδιαφερόμαστε εδώ στην αίθουσα να έχουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορία ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτού οι οποίοι ε, ταξιδεύουν με κάποια πτήση αλλά και για αυτού οι οποίοι ε, ζουν σε περιοχές τις οποίες περνούν από πάνω αεροπλάνα. Θέλουμε λοιπόν επίσης να έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ε, ε, ε σε, για το περιβάλλον και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Πέραν λοιπόν του υψηλού επίπεδου ασφαλείας ε, της αεροπορίας παρέχουμε και κάποιες άμεσες υπηρεσίες στον κλάδο και γι' αυτό ακριβώ και έχουμε μεικτή χρηματοδότηση και παρέχουμε υπηρεσίες μέσω μιας ενιαίας ε, ε, διαδικασίας ε, κανονισμού και πιστοποίησης, κάτι το οποίο επιτρέπει να έχουμε ενοποιημένα στοιχεία στον κλάδο και φυσικά διευκολύνουμε και την ενιαία αγορά εσωτερικής αεροπορίας προκειμένου να διευκολύνουμε και τους τρόπους με τους οποίους ο κλάδος της αεροπορίας μπορεί να δραστηριοποιείται. Υπάρχει τέλος και μια ακόμα πτυχή στην αποστολή του οργανισμού να να δούμε την ανάπτυξη και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, κυρίως με άλλους οργανισμούς αεροπορίας και άλλους ρυθμιστές, την ΑΙΚΑΟ και άλλους φυσικά ε, που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι η Άσα δεν δραστηριοποιείται αυτόνομα, αλλά ε, δημιουργούμε ένα σύστημα εταιρικών σχέσεων. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά με εθνικές αρχές, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για τη δημιουργία ενός ε, συστήματος αεροπορίας και η ΆΣΑ δεν εργάζεται αυτόνομα, ανήκουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο προσπαθούμε και να προωθήσουμε. Εάν τώρα περάσουμε στις πτυχές του προπολογισμού. Ο νομοθέτης, ή μάλλον να το παραλλιώσω. Να ξεκινήσουμε από τον προπολογισμό. Έχουμε ένα προπολογισμό περίπου 142 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και από ό,τι βλέπετε ε, ο ΕΑΣΑ χρηματοδοτείται από τρεις βασικές πηγές. Ο πρώτος οι υπηρεσίε που παρέχουμε στον κλάδο για τον οποίο ε, χρεώνουμε ε, τέλη ή αμοιβέ ανάλογα από την υπηρεσία που προσφέρεται και αυτό ε, αντιστοιχεί σε 96 ε, εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η δεύτερη πτυχή είναι ρυθμιστικές δραστηριότητε της Ένωσης, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ενισχύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεισφορά των άλλων κρατών μελών, περίπου 39 εκατομμύρια. Και επίσης υπάρχει πλέον από εδώ και 2-3 χρόνια όλο ένα και πιο μεγάλη χρηματοδότηση για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη διεθνή τεχνική συνεργασία μέσω συγκεκριμένων δημοσιονομικών μέσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω ε, τι συνθήκε ε, παγόδα ή ε, από τον τομέα της έρευνας τον ορίζοντα 2020. συμμετέχουμε πλήρως σε τέτοια προγράμματα. Άρα έχουμε τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης τελικά στον ΕΑΣΑ. Τώρα, πώς διαχειριζόμαστε αυτόν τον προπολογισμό. Όπως ε, ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς εφαρμόζουμε το λεγόμενο μοντέλο ανάθεσης εσόδων, assigned revenue ο νομοθέτης στο βασικό κανονισμό, στο άρθρο 65, προβλέπει σαφώς ότι τα τέλη και οι αμοιβέ οι οποίες καταβάλλονται από τον κλάδο θεωρούνται ε, τέτοια μορφή έσοδα. Υπάρχει λοιπόν η νομική υποχρέωση για μας να εφαρμόζουμε αυτό το μοντέλο και ε, μπορεί να σας φαίνεται πολύ τεχνικό αλλά η ιδέα είναι πολύ απλή. Τα έσοδα από αυτές τις αμοιβέ και τα τέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο. Δηλαδή, ο κλάδος που καταβάλει τα ποσά αυτά για τις πληρωμές θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά τα οποία καταβάλλονται χρησιμοποιούνται μόνο για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει διασταυρούμενη ενίσχυση μεταξύ των διαφορών ε, πηγών χρηματοδότησης και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να ε, μπλέξουμε τις τρεις κατηγορίες ε, χρηματοδότησης που έχουμε. Πρέπει να δαπανούμε για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Αυτό το μοντέλο ε, έχει και κάποιους περιορισμούς μεν, αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό. Και πώς τα διαχειριζόμαστε. Υπάρχει ένα μοντέλο λογιστικού κόστους που βασίζεται στα υψηλότερα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ό,τι δηλαδή εφαρμόζουν όλες οι μεγάλες ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και βασίζεται και στην εφαρμογή ε, ε, ε ενός συστήματος ERP, το οποίο είναι το SAP, το SAP που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία, το οποίο ελέγχεται και από εξωτερικούς ελεγκτές γιατί είναι τμήμα του, ενιαίου, ε, του ετήσιου ελέγχου του οργανισμού. Αυτός ο ξεκάθαρος διαχωρισμός που ανέφερα ε, βασίζεται στον ε, οριζόντιο κανονισμό, αλλά είναι και μέλημα του κλάδου. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι οτιδήποτε καταβάλουν στον οργανισμό δίνεται μόνο για δραστηριότητες πιστοποίησης. Κατά συνέπεια, μεταφέρονται ποσά από τη μια χρονιά στην άλλη και το πλεόνασμα το οποίο μπορεί να έχουμε από τις δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, δηλαδή και τις χρεώσεις και τις αμοιβέ ε, και ε, τα λεφτά τα οποία δίνονται για τα προγράμματα, ε, διατηρείται προκειμένου να ε, δαπανηθεί τις επόμενες χρονιές ή να χρησιμοποιηθεί για ε, ισοζύγιο τυχών μελλοντικών ζημιών. Στο θέμα της ενίσχυσης, το πλεόνασμα επιστρέφεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το πλεόνασμα όμως το οποίο έχουμε από την πλευρά της ενίσχυσης, που σημαίνει ότι ο οργανισμός ε, έχει πολύ μεγάλες μεταφορές ποσών και ε, συσσωρευμένο πλεόνασμα, αλλά αυτό είναι τμήμα του προϋπολογισμού, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τις επόμενες χρονιές. Λοιπόν, το σύστημα είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένε δράσει, ε, τι οποίε ανατίθεται συγκεκριμένα κονδύλια ε, για ό,τι ακριβώ γίνεται. Άρα είναι αντιπροσωπευτικό και σημαίνει ότι χρειάζεται και κάποια ε, διαφάνεια και αυτή την προσδοκία έχουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιος ο κλάδος αλλά είναι και σύνθετο. Είναι πολύ πιο σύνθετο από το ενιαίο μοντέλο το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πιο σύνθετο διότι δεν υπάρχει καμία ευελιξία μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης και πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική διαχείριση ε, στη διάρκεια της χρονιάς ε, ε, για την επανάληψη μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης και η επανάληψη στο σύστημα των λογιστικών είναι πολύ περίπλοκη, διότι βασίζεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιο έχει προγραμματίσει να δραστηριοποιηθεί σε μία από τι τρει δραστηριότητε και είναι σε άλλη, τότε το σύστημα θα λάβει υπόψη του αυτή τη συγκεκριμένη δαπάνη. Ο καταμερισμό δηλαδή μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυναμικό και εξαρτάται από τι διάφορε δραστηριότητε και εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το προσωπικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η υποβολή εκθέσεων είναι πιο ε, περίπλοκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ορισμένες φορές και λίγο πιο δύσκολες, διότι πρέπει να λάβουμε σαφώς υπόψη και τον καταμερισμό μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Φέτος, για παράδειγμα, είχαμε απώλεια ζημίες στο θέμα των ενισχύσεων, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε όμως αυτό αυτή τη ζημία που έχουμε στην ενίσχυση να την ισοσταθμίσουμε από το ποσό που έχουμε στις αμοιβέ, πρέπει να περιμένουμε και να το λάβουμε υπόψη μας στον επόμενο προπολογισμό. Και αυτό σημαίνει ότι οποιασδήποτε σημαντικές επενδύσεις οι οποίες αφορούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν όπως ε, θα γινόταν στο ενιαίο μοντέλο γιατί υπάρχει χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές. Πρέπει τα ποσά λοιπόν να είναι διαθέσιμα βάσει των συγκεκριμένων ποινών. Αν έχουμε λοιπόν μια σημαντική επένδυση που αφορά ευρωπαϊκή ενίσχυση είναι πολύ ε, λιγότερη ευελιξία από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στις ε, αμοιβέ και στα τέλη. Στη συνέχεια, γίνεται πλήρης διαχείριση του προϋπολογισμού βάσει των συγκεκριμένων γραμμών προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και το θέμα της αποτελεσματικότητας. Αναφέραμε αυτή την πιλωτική ε, διαδικασία στην οποία μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις προσπαθούμε να καθορίσουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα το φόρτο εργασίας του οργανισμού και συνεργαζόμαστε στενά και με τον κλάδο της αεροπορίας, αλλά επιπλέον, και αυτό είναι και άλλο τμήμα του πιλωτικού προγράμματος, ε, στη ΝΕΑΣΑ έχουμε εφαρμόσει ένα ε, πρόγραμμα το οποίο εξετάζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για να μπορούμε να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά και να έχουμε και κάποια ωφέλη όπως ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα 2% περιθώριο, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μόνο όταν υπερβούμε αυτό το 2% αρχίζει να έρχεται επιπλέον χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν και νέα ε, μοντέλα, τα οποία ε, τα αναθεωρούμε με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δεύτερο τμήμα του πίνακα βλέπετε ότι ο οργανισμός αύξησε και το προσωπικό ε, το οποίο χρησιμοποιούσε για επιχειρησιακές δραστηριότητες. Πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει πολύ μεγάλη επιρρογνωμοσύνη. Το 81% του προσωπικού ε, απασχολείται σε ε, επιχειρησιακά καθήκοντα και αν λάβουμε υπόψη το γεγονός αυτό και το ότι υπάρχει ένα ορόσημο για συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο ασχολείται με διοικητικές ε, διαδικασίες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το ενιαίο μοντέλο έχει πολύ λιγότερο γραφειοκρατικό άχθο. Ε, νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε μόνοι σα συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία τα οποία σα δίνουν, λαμβάνοντα υπόψη και το πόσο περίπλοκο είναι να διαχειρίζεται κανεί διαφορετικέ πηγέ χρηματοδότησης. Η κατάσταση του ΕΑΣΑ αυτή τη στιγμή ε, είναι ε, αρκετά καλή οι δείκτες ε, για τους χρηματοοικονομικούς πόρους είναι αρκετά υψηλοί. Έχουμε ε, υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού ε, και το υψηλότερο που είχαμε ποτέ και έχουμε και πλήρη χρήση όλων των θέσεων που σημαίνει ότι ο ΕΑΣΑ έχει προσλάβει όλους τους υπαλλήλους που προβλέπονται βάσει προπολογισμού στον οργανισμό. Ε, με τα χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω, ε, κύριε Μάστιο, ότι ε, το ε, σχέδιο ε, της ΕΑΣΑ πραγματικά ενθαρρύνει τους οργανισμούς ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τη χρηματοδότηση των οργανισμών τους από ό,τι κάνουν στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε με την Κομισιόν και το θάρρος να δοκιμάσουμε ένα μοντέλο το οποίο έχει καλές δυνατότητες να εφαρμοστεί και σε άλλες ε, και σε άλλους οργανισμούς ε, θα πρέπει να προσαρμοστεί μεμονωμένα, όμως πιστεύω ότι ε, κάθε κράτος μέλος μπορεί να κερδίσει από όλο αυτό ε, δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, έχουμε ανεξέλεγκτες, ανεξέλεγκτες συνέπειες με βάση τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην αποτελεσματικότητα, να προσαρμόζονται οι έλεγχοι του προπολογισμού με βάση τις ανάγκες της αγοράς και ταυτόχρονα έχουμε βρει έναν πολύ καλό τρόπο, ο οποίος χρηματοδοτείται και καλά ε, και δεν επηρεάζει τα κράτη-μέλη ε, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Επίσης ε, έχουμε μαζί μας όπως προαναφέρθηκε το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σάτσιος αν θα ήθελε να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως ε, το ε, θέμα το οποίο συζητάτε αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου σε αυτό το εργαστήρι είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και για εμένα προσωπικά διότι είμαι μέλος του, της ομάδας ελέγχου των οργανισμών βέβαια δεν, είμαι, δεν έχω προετοιμαστεί ούτως ώστε να κάνω μια ε, συγκεκριμένη ε, έκθεση σχετικά με τα όσα παρουσίασε η κυρία ε, Βος. Παρόλα αυτά όμως θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας κάποιες σημειώσεις που έχω κάνει οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στον διάλογο. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι εφόσον εκπροσωπώ το ελεγκτικό συνέδριο έχουμε ε, ισχυρές αλλά περιορισμένες εξουσίες και γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα να περιοριστώ σε ζητήματα τα οποία αφορούν την ορθή διαχείριση των, ε, των πόρων είναι έργο των ε, νομοθετών, ε, των ε, μελών του Κοινοβουλίου να κάνουν τον, τον έλεγχο των οικονομικών παρόλο αυτό όσον αφορά την ορθή διαχείριση των δημοσιονομικών το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να κάνω είναι να συστηματοποιήσω τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς που είναι πλήρως ή μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενοι. Έκανα μία λίστα λοιπόν 10 συνολικά οργανισμών, δεν είναι όπως παρουσίασε η Κομισιόν είναι δύο παραπάνω. 10 ε, ε, λοιπόν οργανισμών ε, που χρηματοδοτούνται μερικώς από τα κράτη-μέλη από, τις ή από τη βιομηχανία. Βρήκα έξι διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης για 10 συνολικά οργανισμούς. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο εύρος χρηματοδότησης, μια μεγάλη ποικιλία χρηματοδότησης, κάτι το οποίο είναι τεράστιο. και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε οργανισμός ε, έχει ε, δημιουργηθεί ε, για συγκεκριμένο σκοπό, για μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική εντόπισα μονάχα δύο οργανισμούς ε, που κατ' εμέ φαίνεται ότι χρηματοδοτούνται με παρόμοιο τρόπο. Ε, πρόκειται για το ε, Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών καθώς επίσης και για, την, και για το EPO. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρόσεξα είναι ότι κανένας οργανισμός ε, δεν έχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο χρηματοδότησης. Ξεκάθαρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτείται ε, ξεκάθαρα ε, από άλλες πηγές και όχι από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Όπως δήλωσε λοιπόν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έχουμε ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά ταμεία αλλά έχουμε και άλλα θέματα όπως είναι τα Ευρωπαϊκά ευρωπαϊκά ε, σχολεία. Αν λοιπόν αρχίσουμε να απαριθμούμε με βάση ε, το ε, κόστος για να σχεδιάσουμε τη χρηματοδότηση και να υπολογίσουμε τις συμβουλές οι οποίες θα πρέπει να συλληφθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα είναι μια απλή, ένας απλός υπολογισμός. Δεν θέλω να διαπαρτηρηθώ όμως είναι πολύπλοκο ε, το γεγονός ότι αυτές, αυτοί οι οργανισμοί που φαίνονται ότι είναι ε, πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενοι εντοπίζεται από το ελεγκτικό συνόδριο ότι τελικά χρηματοδοτούνται και από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο, αποτελεί υποχρέωση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου με βάση τις συνθήκες, όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό επιτέλους ε, να ε, συμμετέχουμε ε, στα αποτελέσματα και στις εκθέσεις όλων αυτών των υπηρεσιών και παρά όλα τα μοντέλα τα οποία εντυπώσαμε όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι οργανισμοί ανήκουν στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό απαιτεί τόσο μια πολιτική προσέγγιση σε όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα και μια προσέγγιση σχετικά με την ορθή ε, διαχείριση των δημοσιονομικών τους. Ε, άλλα ε, τέσσερα ζητήματα, τέσσερις αρχές τις οποίες θα ήθελα να τονίσω συγκεκριμένα είναι οι εξή. Πρώτον, έχουμε διαφορετικά επιχειρησιακά μοντέλα ε, modus operandi ε, των ε, οργανισμών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα για τους οργανισμούς, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει ένα σωστό κίνητρο για να ξοδευθούν μεγάλα ποσά ε, για ε, τα ε, αποθεματικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί τότε όλο αυτό δεν πρόκειται να συμφωνεί με την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Βέβαια όλο αυτό μπορεί να έχει και πολιτικές συνέπειες ε, σε περίπτωση ε, που Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι πολίτες ε, παρατηρήσουν ότι κάποιο ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμός άρχιζε απλά να δαπανά χρήματα τότε αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ πιο δυσάρεστες συνέπειες από την ίδια τη δαπάνη των χρημάτων. Το άλλο θέμα αφορά τη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι η αρχή η οποία ε, πιστεύω ε, είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να επενδύσουμε δημόσια χρήματα. Ε, κοστίζει αλλά αξίζει το κόστος για τον λόγο τον οποίο μόλις ανέφερα για τους Ευρωπαίους πολίτες και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το οποίο επίσης ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση αλλά και από την άποψη της αρχής ε, των ε, του ορθού προϋπολογισμού δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, ξεκάθαρο το ζήτημα του προϋπολογισμού. Μιλήσαμε για τις μεταφορές ποσών τονίσαμε ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, λύσεις ε, ε, για τις μεταφορές όμως εγώ πιστεύω ότι αναλογικά το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα αποθεματικά των αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών διότι και εκεί πρόκειται για ένα είδος μεταφορών όπως τονίστηκε σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε κάποιες ε, γενικές αρχές ε, οι οποίες ε, θα οδηγήσουν και σε καλύτερη ποιότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Και τέλος όσον αφορά την λογοδοσία και τη δημοκρατική επίβλεψη ακριβώς για τους λόγους τους οποίους ανέφερα προλίγου πιστεύω ότι η πλήρωση μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί ε, ή οποιοδήποτε οργανισμός ε, θα πρέπει να υπόκειται ε, σε δημοκρατική επίβλεψη και εποπτεία θα πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες διαδικασίες όπως συμβαίνει σε αυτές οι οποίες χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν θεωρεί ότι ε, κάποιο είδος ε, διαδικασίας απαλλαγής θα πρέπει να υπάρχει για αυτές ε, τις υπηρεσίες ε, διότι ανήκουν ε, σε αυτό το ε, σύνολο οργανισμών που χρησιμοποιούν τους κανονισμούς για τη λειτουργία των θεσμών της Ένωσης και θα ήταν ορθό να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω τις απόψεις μου. Ευχαριστούμε και εμείς για τις δηλώσεις σας διότι με βάση αυτό δεν γνώρισα ότι έχουμε 10 οργανισμούς που ακολουθούν εντελώς διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης. Ε, θεωρούσα ότι υπήρχαν κάποιες βασικές ε, ομοιότητες, όμως τελικά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές στα συστήματα που θα πρέπει να τις ξεπεράσουμε όσον αφορά τις δικές μας επιτροπές. Εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα για να το εξετάσουμε και να δούμε ιστορικά πώς φτάσαμε σε αυτό ε, το σημείο πώς εξελίχθηκε ε, η κατάσταση, ε, οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούνταν σε διάφορες χρονικές περιόδους, με διαφορετικούς στόχους, με αποτέλεσμα κάθε οργανισμός να έχει διαφορετικούς στόχους. Το γεγονός ότι έχουμε τόσους πολλούς οργανισμούς, το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις δικές μας επιτροπές, διότι θα θέλουμε να έχουμε μια βάση, μια δυνατότητα, ούτως ώστε να υπάρχει μια εποπτεία πάνω σε όλο αυτό ε, και είναι σημαντικό το γεγονός ότι αναφέρθηκε όλο αυτό και ότι εφόσον ακόμα και στην περίπτωση μιας πλήρους χρηματοδοτούμενης υπηρεσίας και οργανισμού θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ε, εποπτείας. Όλο αυτό έχει να κάνει με το ε, γεγονός ότι ε, εξυπηρετεί ε, τους πολίτες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Θα ήθελα αρχικά να δώσω το λόγο στα μέλη. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, παρακαλώ πείτε το μου. Ευχαριστώ. Θα κάνω ορισμένα καταληκτικά σχόλια και στο τέλος, αλλά είχα ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένα, το οποίο μάλλον θα απευθύνω στους οργανισμούς. Αφορά το θέμα της εποπτείας και των απαλλαγών. Καταλαβαίνω γιατί οι οργανισμοί θεωρούν ότι η διαδικασία των απαλλαγών και η εμπλοκή του Κοινοβουλίου δεν είναι κάτι το ευκταίο γιατί ε, χρηματοδοτήστε πλήρωση εν μέρη από αμοιβέ. Όμως όπως είπαν και άλλοι υπάρχει και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ε, συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και νόμους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια, κάποιος δημοκρατικός έλεγχος. Κύριε Εκφαρτ, στα τέλη της παρουσίασής σας αναγνωρίστε τουλάχιστον εν μέρη αυτή την αρχή και είπατε ότι είστε θετικά διακείμενος σε, σε ορισμένες συζητήσεις για μελλοντική συνεργασία με το Κοινοβούλιο μπορείτε να σταθείτε λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα. Εννοείται δηλαδή ότι μία φορά το χρόνο οι οργανισμοί θα έρχονται δηλαδή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, θα μας κάνουν μια παρουσίαση και θα συζητούν μαζί μας. Θα ήσασταν διατεθειμένος να κάνετε κάτι τέτοιο ή να κάνετε κάτι άλλο που να ακολουθεί την άγουσα της συνεργασίας. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όταν γίνεται λόγος για μη εποπτεία, είπα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και ε, μας ελέγχει το ελεκτρικό Συνέδριο και ο κλάδος που πληρώνει ε, μας ελέγχει προσεκτικά στέλνουμε όλα τα έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημοσιεύουμε τα πάντα στον ιστότοπό μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει ε, τέτοια δημοκρατική εποπτεία. Εάν τώρα το Κοινοβούλιο θα ήθελε κάτι παραπάνω, δεν το αποκλείω. Γιατί όχι. Να έρθουμε και να σας ε, παρουσιάσουμε όποια στοιχεία επιθυμείτε. Κανένα πρόβλημα. Να το κάνουμε αυτό μια φορά το χρόνο. Βέβαια, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό θα πρέπει να αλλάξει και ο ιδρυτικός μας κανονισμός. Ε, έχει τροποποιηθεί τώρα ε, πρόσφατα ο ιδρυτικός κανονισμός του EUIPO, αλλά βεβαίως με τα χαράς να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο πιθανούς τρόπους ε, συνεργασίας. για να δηλώνετε και εσείς ικανοποιημένοι από τις εργασίες ε, του οργανισμού μας και για να ε, καλύπτονται και ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως, μπορούμε να το εξετάσουμε στο μέλλον αυτό. Τόμας, δεν ξέρω ποιος ζήτησε πρώτος το λόγο. Είσαι ευγενικό, πάντα το έλεγα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρουσιάσεις σας μας παρουσιάσετε ε, τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών σας. Προς τον κύριο Σιλβάνο Πρέζα μιλήσατε για το αποθεματικό, το πλεόνασμα μάλλον ε, ε, των οργανισμών όταν έχουμε μεταφορά πόρων στον επόμενο προπολογισμό. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο υπάρχει ένα προκαθορισμένο ποσοστό για αυτά τα ποσά Εάν δεν έχει προκαθοριστεί το ποσοστό, μήπως θα έπρεπε να το καθορίσουμε. Και μία σκέψη ακόμα. Εάν ε, περισσεύουν πόροι και μπορούν να θεωρηθούν πλεόνασμα, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει πλεόνασμα. Μήπως επειδή οι οργανισμοί δεν έχουν ε, υλοποιήσει το πρόγραμμά τους πλήρως, υπάρχουν άλλοι λόγοι και την επόμενη χρονιά ο οργανισμός λαμβάνει νέους πόρους. Διερωτώ με λοιπόν κατά πόσο αυτό λειτουργεί αθρηστικά. Έχετε άλλα στοιχεία. για το μέγεθος αυτών των μεταφορών ποσών σε σχέση με το συνολικό εισόδημα ενός οργανισμού. Ευχαριστώ. Τόμας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την εξαιρετική αυτή συζήτηση. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για απαλλαγές ε, ευρωπαϊκών οργανισμών πολλές φορές και έτσι πολλές φορές έχω επισκεφτεί τέτοιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και πραγματικά τα όσα αναφέρθηκαν να βρίσκουν σύμφωνο. Θεωρώ ότι ω μέλη της, ε, των, των Επιτροπών Προπολογισμών και Ελέγχου του Προπολογισμού πρέπει να λειτουργούμε πολύ συστηματικά και να εξετάζουμε τι λειτουργίε και τι ενέργειε ε, αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι περισσότεροι έχουν μόνο ε, μερική πληροφόρηση για αυτούς τους οργανισμούς. Περισσότεροι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν καν ότι οι οργανισμοί εδρεύουν ε, στις χώρες τους. Για παράδειγμα, ξέρω ότι ε, ο διαστημικός οργανισμός είναι στην Πράγα. Πολλοί συνάδελφοί μου όμως δεν το ήξεραν. παρότι είναι τεράστιες εγκαταστάσεις του οργανισμού αυτού στην Πράγα. Όμως ε, η προβολή είναι ελλειπής. Επομένως, πρέπει να έχουμε λοιπόν μία εποπτεία των οργανισμών. Αν δείτε τους φακέλους απαλλαγών για κάθε οργανισμό, έχουμε έναν φάκελο για σας. Όταν υπάρχει πρόβλημα στον τύπο, ε, το αρχιοθετούμε. Μπαίνει δηλαδή στο φάκελό σα. Και κατά τη διάρκεια των απαλλαγών ε, προσπαθούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί σα. Κάποιε φορέ είναι ίσονο σημασία. Αλλά, για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδε πήγα στη Βιέννη. Και συζήτησα ένα θέμα που αφορούσε το προσωπικό με κάποιον και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ένας από τους ε, πρώην υπαλλήλους σας ήρθε σε επαφή μαζί μου για να συζητήσει ένα τέτοιο θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, είναι αποτελεσματικός εδώ ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούν όλοι οι οργανισμοί ε, να χρηματοδοτούνται από αμοιβέ. Σε παράδειγμα, η Europol από ποιον ας πούμε, θα καταβάλλονται αυτέ οι αμοιβέ. Για κάθε εγκληματία δηλαδή που πιάνουμε και ε, για κάθε κατάσχεση ας πούμε, παράνομων εμπορευμάτων παίρνουμε ένα ποσοστό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά οι αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί, όπως ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ε, κάποιες διασυνδέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινοβουλίου και όσων επιχειρήσεων λαμβάνουν αυτές τις άδειες, όπως Boeing, Boeing Airbus κτλ. Συχνά έχω μιλήσει για αυτές τις δύο εταιρείε και βλέπω ότι όταν κανείς ε, αναφέρει την ΙΑΖΑ είναι μια σφραγίδα ποιότητας, αν θέλετε. Είναι σαν ένα τέτοιο σήμα ποιότητας και ασφάλειας. όλη αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο ε, τα οικονομικά ζητήματα. Είναι και θέμα ποιότητας και ασφάλειας. Και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι ακριβώς μια εγγύηση ποιότητας. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θεωρώ ότι και πάλι υπάρχει περιθώριο εξοικονόμησης πόρων. Για παράδειγμα, υπήρχε μία ε, συνεδρίαση μιας ημέρας ε, στη Βουδαπέστη ε, με τη ΣΥΠΟΛ και συμφωνήσαμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερη ε, διάθεση των προσλήψεων, καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων, καλύτερη διοργάνωση των διαγωνισμών. Κατανοώ ότι οι ανάγκε τη ΕΠΟΛ και τη CIT διαφέρουν. Όμω πρέπει να βρούμε τρόπου να έχουμε, για παράδειγμα, κοινού διαγωνισμού ό,τι αφορά του ε, υπολογιστέ ή ορισμένε υπηρεσίε. Γιατί οι οργανισμοί βρίσκονται και κοντά. Επομένω μπορούμε έτσι να εξοικονομήσουμε πολλού πόρου. Κάτι τελευταίο, συνάδελφοι. Ήμουν ε, αρμόδιος για την απαλλαγή ορισμένων ευρωπαϊκών οργανισμών το 2014 Και πραγματικά ήθελα να βρω λάθη. Και να σας ε, διδάξω, ένα, να σας δώσω ένα μάθημα, για να θέλετε, στο πλαίσιο της απαλλαγής. Αλλά πραγματικά η ποιότητα της δουλειάς σας έχει αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια που δεν είχαμε και πολλά για να σας κατακρίνουμε. Μπορούμε μόνο να σας ενθαρρύνουμε να βρείτε νέο κίνητρο για να βελτιώσετε και να προωθήσετε το έργο σας. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική σας αδυναμία. Δεν μπορείτε να προβάλλετε το πόσο καλοί είστε. Και αν το κάνετε αυτό θα είχαμε 150 ακροάσεις και εργαστήρια για τους τρόπους χρηματοδότησής σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να σας ε, ε, εξετάζουμε και να σας ανακρίνουμε για το πώς διαχειρίζετε τα κονδύλια σας. Αλλά εκεί δεν βρίσκουμε λάθος. Όμως πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε το έργο σας και προς τα εμάς και προς άλλους, αλλιώς θα υπάρχει πάντα δυσκολία. Στην τελευταία οριζόντια απαλλαγή δώσαμε την ευκαιρία να αυξήσετε το προσωπικό σας συνολικά σε όλους τους οργανισμούς. Παρακαλώ, αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα. για να προβάλλετε το έργο σας σε εμάς, στο Κοινοβούλιο και στους Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Νομίζω ήταν σημαντικό αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους να απαντήσουν στα σημεία αυτά και στις ερωτήσεις. Δεν ξέρω σε ποιον απευθυνόσασταν ακριβώ, αλλά νομίζω ότι μία απευθυνόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σω θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση τη κυρία Σουλίν και το, προς, προς το δικτύο θα μπορούσε να απαντήσει την ερώτηση του Τόμας ε, για την περαιτέρω αυξημένη συνεργασία, για την ε, πρόσκληση σε διαγωνισμούς, ε, προσλήψεις κλπ. Αν οποιοδήποτε άλλος όμως θέλει να απαντήσει, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Βον. Όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Σουλίν, για τη μεταφορά των πλεονισμάτων. Ε, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μερίδιο το οποίο καθορίζεται. Ε, κάνουμε διάκριση μεταξύ των οργανισμών τα, οι οποίοι είναι πλήρως ε, ε, αυτοχρηματοδοτούμενοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Για τους πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους ε, στην πραγματικότητα είναι και εκτός πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας του ευρωπαϊκού προπολογισμού, διότι δεν συμπεριλαμβάνονται καν στον προπολογισμό και επομένως από εκεί και πέρα επαφίεται στην ε, ίδια τη δομή της διακυβέρνησης των οργανισμών. Υπάρχει για παράδειγμα το παράδειγμα του ε, γραφείου ε, των φοιτικών ποικιλιών. Ήδη από τα όσα χρεώνουν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση. Υπάρχει λοιπόν ένα ενσωματωμένο σύστημα διακυβέρνησης το οποίο προσαρμόζει το επίπεδο των πλεονασμάτων και του αποθεματικού ε, και υπάρχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει η άλλη περίπτωση του ΆΙΠΟ στο Αλικάντε, όπου υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πλεόνασμα, το οποίο συσσωρεύεται σύν το χρόνο, και νομίζω ότι είναι πάνω από 450, 400 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει σύστημα το οποίο ε, επιτρέπει την απόσβεσή του. Ε, πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες βεβαίως του κάθε οργανισμού, αλλά υπάρχει το θέμα αυτό για τους άλλους οργανισμούς που εν μέρη αυτοχρηματοδοτούνται και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται ε, από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, υπάρχει μια διαδικασία προσαρμογής στον ετήσιο προπολογισμό. Όταν υπάρχει πλεόνοσμα, λαμβάνεται υπόψη για να δούμε και τις ανάγκες για ε, ε, φρέσκο χρήμα, όπως το αποκαλούμε, για την επόμενη χρονιά. Επομένως, προβλέπεται ένα πλεόνασμα το οποίο ε, χρησιμοποιείται για να καλύψει τμήμα των δαπανών και από εκεί και πέρα δίνεται και έγκριση για νέες δεσμεύσεις υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλεόνασμα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία προσαρμογής, η οποία είναι ενσωματωμένη ε, στην ετήσια δημοσιονομική διαδικασία. Για τα ποσά ε, προτείνω να σας στείλουμε γραπτός ε, τα στοιχεία γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ε, γνωρίζω επακριβώς τα ποσά των πλεονασμάτων. Μπορούμε να στείλουμε τον πίνακα όμως στη γραμματεία της Επιτροπής και να σας δοθεί αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Σπανιόλη. Ναι, ευχαριστώ. Πράγματα. Ο τομέας των κοινών ε, προσκλήσεων υποβολής προσφορών ε, φέτος ε, και με την Προεδρία μας, αλλά θα συνεχιστεί στο μέλλον αυτό. Στην επόμενη συνεδρίαση θα επισημοποιήσουμε την σύσταση ενός επίσημου υποδικτύου για του διαγωνισμούς των οργανισμών και μαζί τους έχουμε ξεκινήσει ένα κοινό πρόγραμμα προσκλήσεων υποβολής προσφορών Υπάρχει μια συγκεκριμένη δικτυακή πύλη για τις δραστηριότητες του δικτύου και πώς θα τις διαχειριζόμαστε εξ ονόματος των οργανισμών και των υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλά ενεξελίξη. Αναφερθήκαμε στην υπηρεσία του cloud ε, που είχαμε πέρσι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Εξετάζουμε πολλά άλλα, αν μπορούμε να κάνουμε μαζί αγορά υπηρεσιών ε, ελεγκτικών, για παράδειγμα, ε, και αίθουσες συνεδριάσεων, εξοπλισμό, προσωρινό προσωπικό, ε, υπηρεσίες κινητής, τηλεφωνίας. Ε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι στα σκαριά και μπορούν να ε, αγοραστούν από κοινό από τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ο πιο πολλά υποσχόμενος τομέας υπηρεσιών που θα μπορούσαμε να έχουμε. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες εργασίες εν εξελίξη και ελπίζουμε να τα βελτιώσουμε στο δυνατόν περισσότερο. Επίσης, να διαβεβαιώσω τον κύριο Ροζόφσκι ότι επεκτείνουμε την μόνιμη γραμματεία του δικτύου στις Βρυξέλλες. Θα αλλάξει και όνομα, θα είναι Shared Support Office, ε, θα στελεχώνεται από περισσότερο προσωπικό. Έχει αναγνωριστεί ήδη η ανάγκη να υπάρχει ε, μια πιο κεντρική, ισχυρή δομή για να διαχειρίζεται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ε, η κοινή δικτυακή πύλη για τους διαγωνισμούς και οι κατάλογοι και κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ε, εποφελεί, δημιουργούν συνέργειες και αποτελεσματικά στοιχεία σε επίπεδο οργανισμών και δικτύου και πρέπει να τα κάνουμε από κοινού σε κεντρικό επίπεδο και πρέπει να υπάρχει και ε, κοινή δομή ε, στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος από τους άλλους ομιλητές ε, το λόγο ή να απαντήσει. Παρακαλώ. Δύο λόγια να πω για το θέμα της έρευνας, ε, από των αποθεματικών, συγγνώμη, γιατί έχουμε αποθεματικά. Ε, για να τα πούμε πρακτικά τα πράγματα. Πρέπει να καθορίζουμε αμοιβέ ε, και σε επίπεδο οι οποίες ε, θα επιτρέπουν να έχουμε και ε, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Βέβαια αυτό είναι αδύνατο γιατί δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος πόσες αιτήσει θα έχουμε. Αν λοιπόν καθορίσει κάποιο τι αμοιβή, δεν μπορούμε να τι αλλάζουμε και κάθε χρόνο. Εμεί η πολιτική μα είναι να τι καθορίζουμε κάθε τέσσερα χρόνια και εδώ και 4-5 χρόνια ε, λειτουργούμε με έλλειμμα στον προπολογισμό προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε το αποθεματικό. Ε, τώρα α, ήρθε η στιγμή, αλλάξαμε τις αμοιβέ για να τα ε, αντιστρέψουμε αυτά για να έχουμε πλεόνασμα και να είμαστε όσο ε, πιο κοντά σε ισοσκελισμένο προπολογισμό. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και το αποθεματικό ε, εξ αρχής το Συμβούλιο ε, του ΣΥΠΙΒΕΟ αποφάσισε ότι το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών θα μπορούσε να είναι ένα σωστό επίπεδο γιατί πρέπει να προβλέψουμε και κάποιες ε, απρόβλεπτες εξελίξεις. Τώρα είμαστε λίγο κάτω από αυτό. Είμαστε περίπου στις 500.000 ευρώ και το 50% θα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν εξηγεί και γιατί υπάρχει το αποθεματικό. Και επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω και με αυτό που είπε ο πρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια. Ε, με αυτό αποφεύγουμε και πολλές ανησυχίες ε, που εξέφρασαν αρκετοί και ε, φυσικά και τις ανεξέλεκτες διαπάνες ε, διότι είναι πολύ ανοιχτά και διάφανα τα πάντα για να αποφύγουμε και επικρίσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και από άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα αίτημα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το EMA. Έχουμε ένα συνάδελφο παρόν εδώ και ε, νομίζω ότι επειδή είστε και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχετε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω και να συμμετέχω και στη συζήτηση. Δεν έχω να προσθέσω και τίποτα καινούριο στην όλη συζήτηση. Να επαναλάβω όμως ε, και κάποια ερωτήματα από διαφορετική πτυχή όσον αφορά το θέμα του αυξημένου φόρτου εργασία και τη μείωση των πόρων. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Φαρμάκων από το 2014 μέχρι το 2018 θα έχει αυξήσει τα έσοδά του και το φόρτο εργασία κατά 40% και ταυτόχρονα οι πόροι μειώνονται ε, βάσει και των περικοπών του 1 με 2%. Αυτοί οι οποίοι καταβάλουν τέλη για τις αιτήσει τους Ορισμένες φορές φτάνουν και το μισό εκατομμύριο και φυσικά ε, περιμένουν να τους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και επομένως ο οργανισμός ουσιαστικά βρίσκεται μεταξύ της εξής δυσκολίας. Ε, αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνεται το φόρτος εργασίας και απ' την άλλη έχουμε μείωση των πόρων και δεν μπορούμε να ε, παρέχουμε σωστά τις υπηρεσίες μας οι υπηρεσίε αυτό που κάνουν βεβαίω και αναφέρθηκε και προηγουμένω, αρχίζουν να εξετάζουν διάφορε μορφέ πόρων. Προσωρινό προσωπικό, εξωτερικέ αναθέσει, ε, συμβάσει κλπ. Ε, υπάρχει λοιπόν μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε αυτή την κατηγορία που σημαίνει χάνεται γνώση, χάνεται εμπειρία, πρέπει να γίνουν νέε προσλήψει και η διαδικασία αυτή δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα και φυσικά υπάρχουν και κάποιε κατηγορίε προσωπικού που βρίσκονται σε ευαίσθητε θέσει, λεπτέ θέσει δεν μπορούμε να του αντικαταστήσουμε με προσωρινό προσωπικό. Παραδείγματο χάρη, επιστημονικέ γνωμοδοτήσει. Ο οργανισμό παρέχει επιστημονικέ γνωμοδοτήσει στα ε, πρώτα στάδια των εξελίξεων τη ιατρική και ε, σύν το χρόνο διπλασιάστηκαν και στην πραγματικότητα θα μπορούσαν και να δεκαπλασιαστούν οι γνωμοδοτήσεις ε, για τα ερευνητικά κέντρα, ερευνητές κλπ. Αλλά χάρη, ε, λόγω συγγνώμη, των ε, περιορισμών που υπάρχουν δεν μπορεί να παρέχει περισσότερες επιστημονικές νομοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή παρέχουμε 500 με 600 τέτοιες νομοδοτήσεις ετησίων. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να φτάσουμε στις 6.000. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα βγαίνουν νέα φάρμακα και θα φτάνουν στους ασθενούς μας σε κάποια χρόνια και αν αυτά τα πολλά υποσχόμενα φάρμακα αναπτυχθούν σημαίνει ότι θα υπάρχει έρευνα και στην Ευρώπη αλλά λόγω της αύξησης του φόρτου εργασίας και της μείωσης των πόρων ε, και της μείωσης του προσωπικού εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες ε, στους ετούντες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του αποθεματικού, αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία. Και πάλι, επειδή εμεί είμαστε σε ένα οργανισμό που βρίσκεται εκτός Ευρωζώνης έχουμε και ένα επιπλέον στοιχείο κινδύνου και ε, διακυμάνσεων, το, ε, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ε, ένα ποσοστό των δαπανών μας ε, είναι σε δαπάνες, συγγνώμη, οι δαπάνες μας είναι σε λίρες, ενώ τα έσοδά μας είναι σε ευρώ, που σημαίνει ότι οι απώλειες σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σημαίνει ότι έχουμε αύξηση ε, στο επίπεδο των δαπανών. Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit φτάσαμε στο 8 με 10%, που σημαίνει 10 εκατομμύρια ε, αλλαγή στα έσοδα περίπου. Αν πάνε οι συναλλαγματικές ισοτιμίες προς την άλλη κατεύθυνση, επειδή δεν έχουμε αποθεματικό, ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αποθεματικό, δεν υπάρχει ε, δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τέτοιο κίνδυνο. Επίσης, ε, ε αναφέρθηκαν προηγουμένως, ε, αιτήσει και φόρτο εργασίας, ο προπολογισμό μας είναι πάνω από 300 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι 1% διαφορετικά στις προβλέψεις μεταφράζεται σε αλλαγή 3 εκατομμύρια. Και αυτό δεν αφορά μόνο ε, τις προβλέψεις, αλλά και την ε, χρονική στιγμή των αιτήσεων. Αν προβλέψουμε λοιπόν ότι θα έχουμε 110 νέες αιτήσει για αρχική αξιολόγηση κάποιων φαρμάκων, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια έγκριση ε, κυκλοφορίας του φαρμάκου. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε μόνο ότι θα έχουμε 110 αιτήσει, αλλά πότε θα γίνουν και αιτήσει στη διάρκεια του έτους. Και τι έγινε, στο 25% των αιτήσεων, είχαμε σωστά προβλέψει τις 110, αλλά το 25% των αιτήσεων έγιναν τον τελευταίο μήνα του έτους, που σημαίνει ότι υπήρχαν έσοδα, τα οποία έσοδα γίνονται στη συνέχεια πλεόνασμα και επομένω διαγράφεται. Άρα ε, ο οργανισμός έχει και δουλειά που μεταφέρει για την επόμενη χρονιά, γιατί ε, για να διεκπαιρεωθεί η αίτηση χρειάζεται ένα χρόνο περίπου, επομένω έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η λεπτή πτυχή της διαχείρισης. Η μείωση του προσωπικού λοιπόν για μας δεν είναι πρακτικός τρόπος να λειτουργήσουμε διότι δεν έχει συνέπειες μόνο για τον οργανισμό αλλά ευρύτερε συνέπειες και για την καινοτομία και για την έρευνα και για τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων αλλά και από την αμυγός ε, ε, δημοσιονομική σκοπιά υπάρχει και το θέμα της πρόβλεψης, το να μην υπάρχει αποθεματικό, το γεγονός ότι υπάρχουν διακυμάνσεις ε, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και πλέον ο οργανισμός δεν έχει δυνατότητα προστασία σε αυτέ τι περιπτώσει. Και όπω είπατε και το Brexit είναι μια επιπλέον πτυχή. Ε, επειδή υπάρχουν πλεονάσματα θα έχουμε ένα αποθεματικό που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχουμε αποθεματικό, θα πρέπει να μεταφέρουμε ε, προπολογισμό, να γίνουν προσλήψεις όταν θα αλλάξει το προσωπικό, αλλά δεν θα έχουμε αμέσω πόρους διαθέσιμους, θα πρέπει να περάσουμε τη διαδικασία του προπολογισμού για να πάρουμε πόρους και αυτό φυσικά θα καθυστερήσει λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχόμαστε λοιπόν ε, καλή επιτυχία. Ε, οπουδήποτε και αν βρεθείτε στο μέλλον, ε, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη διαδικασία για εσάς και για την υπηρεσία σας. Άλλα σχόλια. Ε, εκπροσωπώ την IPO στις Βρυξέλλες. Ε, αρχικά όσον αφορά την ε, λογοδοσία θα ήθελα να τονίσω όπως είπε και ο κύριος Σέκβατ ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση του κανονισμού χρηματοδότησης σημαίνει ότι έχουμε έναν πρόσωπο του Κοινοβουλίου στο Διοικητικό μας Συμβούλιο το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ευρωβουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο το Ευρωκοινοβούλιο και είναι υπεύθυνοι και για την διαδικασία απελαγής. Τώρα όσον αφορά τις αμοιβέ, αυτό διαφέρει όπως ε, δήλωσε προλίγου ε, και το ελεγκτικό συνέδριο. Στην περίπτωση μας λοιπόν ε, οι αμοιβέ ορίζονται με τον, στον κανονισμό χρηματοδότησής μας όπου αποφασίζουμε το ποσό των αμοιβών. Για να έχουμε λοιπόν μια διαφοροποίηση αυτών των αμοιβών επιστρέφουμε στον νομοθέτη. Τώρα όσον αφορά το πλεόνασμα ισχύει ότι έχουμε ένα ε, πολύ μεγάλο πλεόνασμα δεν είναι 400 ε, ε, όπως προϋπόθηκε αλλά είναι στα 200 εκατομμύρια διότι ο κανονισμός ορίζει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα θα πρέπει να έχουμε ένα, ένα πλεόνασμα το οποίο όμως δεν είναι όλο διαθέσιμο σε εμάς κάποιος άλλος. Ε, θα ήθελε λοιπόν να κάνω τα τελικά μου σχόλια διότι ε, δεν θα ήταν ωραίο ε, να επιστρέψει η κυρία Μάιερ και να είναι άδεια η αίθουσα. Ο συζητήσαμε εδώ κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να μας βοηθήσουν και για το μέλλον. Όσον αφορά το ε, πλεόνασμα, εξετάσαμε ε, το αν θα το, ε, διαθέτει, θα το κρατάει ο ίδιος ο οργανισμός, ούτως ώστε να μειώνει τις αμοιβέ ή να έχει αποδεματικό. Η άλλη ιδέα είναι τα χρήματα αυτά να μεταφέρονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Βέβαια υπάρχει ένα δισταγμό για όλο αυτό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω συζητήσει πάνω σε αυτό. Είχαμε και την πρόταση του ελεκτικού ε, συνεδρίου ε, για τι ε, μεταφορέ και να υπάρχει ένα αποθεματικό αυτών για μελλοντικέ δαπάνε. τώρα σχετικά με το αν οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν περικοπές προσωπικού είδαμε ότι ε, κρατούν το προσωπικό μόνο στο 1,8 ε, για τις ίδιες. Ε, είδαμε το πιλωτικό πρόγραμμα της ΕΑΣΑ, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, διότι θέλουμε να προσφέρουμε ευελιξία στους οργανισμούς αυτούς, διότι ξέρουμε ότι έχουν διαφορετικές ανάγκες από άποψη χρηματοδότησης, προσωπικού και πόρων. Όσο λοιπόν ε, περισσότερη ευελιξία έχουν τόσο το καλύτερο ε, και ε, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα είναι επιτυχές τότε στη συνέχεια η Κομισιόν θα μπορούσε να εξετάσει αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο και σε άλλους οργανισμούς όμως όσον αφορά τώρα την εποπτεία και τις απαλλαγέ εκεί είπατε ε, κάποια ορθά πράγματα. Ε, είπατε ότι ε, έχετε ελέγχους από το ελεγκτικό συνέδριο και αναφέρθηκε και ο ένας οργανισμός όπου συμμετέχουν μέλη του Κοινοβουλίου αλλά πρόκειται για μέλη από την Επιτροπή Γιούρη και όχι από την ΠΑΤΣ και από την Κοντ ε, και γι' αυτό το λόγο και εμείς ε, θα θέλουμε να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις σχετικά με την υποπτία του προϋπολογισμού. Κάτι τέτοιο θα, θα απαιτούσε αλλαγές στον κανονισμό. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια ετήσια συζήτηση σχετικά με τους οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από αμοιβέ μεταξύ αυτών και των επιτροπών μας ε, πιστεύω ότι υπάρχουν λοιπόν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε μια κάποια ε, πρόοδο ε, με την γραμματεία. Θα, η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας πάνω σε αυτό και κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω. Σας ευχαριστώ καταρχάς όλους που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Ε, δεν έχουμε ε, απαντήσεις για όλο, όμως έχουμε μια ξεκαθαρή εικόνα σχετικά με, ε, το πώς έχει η κατάσταση και ίσως στο μέλλον θα μπορέσουμε να βρούμε, να μπορέσουμε να βρούμε απαντήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία το, της Επιτροπής μας που βοήθησε στην διοργάνωση αυτού του εργαστηρίου. Ε, επίσης ε, όσον αφορά τα όσα είπε ο συνάδελφος Τόμας, ε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απαλλαγή του 14, δεν μπορούμε να θα το επαναλάβουμε και φέτος. Οι, οι οργανισμοί αυτοί είναι πολύ χρήσιμοι, κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο για τους πολίτες της Ένωσης, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, παρέχουν υπηρεσίες για τους πολίτες και ταυτόχρονα μας δείχνουν ότι τα ζητήματα ελέγχου του προϋπολογισμού ε, είναι ένα ζήτημα και κάνετε πολύ καλό έργο πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για ε, το έργο σας και ευχαριστούμε και πάλι ε, που ήρθατε εδώ και συνεισφέρατε στο εργαστήρι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. I'm με κάλεσαν τώρα να ε, κάνω τα τελικά ε, σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που ήσασταν εδώ και σας εύχομαι μια καλή ημέρα.